Possiamo Μπορούμε να ξεκινήσουμε τις εργασίες της ημέρας, ε, τις ημέρας που θα είναι πολύ εντατικές εργασίες. Θα, θα εργαστούμε πολύ. Θα πρέπει να είμαστε πολύ... Έχουμε στοχευμένες παρεμβάσεις. Για νόμους νομικούς πρέπει να σας πω Μέσω διαδικτύου θα υπάρχει ε, μετάδοση της συνεδρίας, το ξέρετε. Η μερίσια διάταξη ε, έχει μοιραστεί Όσοι ήθιστε. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θεωρείται συγκεκριμένοι. Θα περιοριστώ να δώσω ελάχιστες ε, ανακοινώσεις για να κερδίσουμε χρόνο. Τα υπόλοιπα θα τα πω στην επόμενη συνεδρίαση. Είναι εδώ ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών της Προεδρίας Ουγγαρίας είναι ο προεδρεύων ε, του Συμβουλίου και θα πρέπει να δώσουμε χρόνο κυρίως εκείνων. Έχω να σας πω τα εξή. Στη συνεδρία της 12 η Ιανουαρίου οι συντονιστές καθόρισαν τους κυρίους Ελμαρ Μπρόκ και Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη σύμφωνα με τη διαδικασία διαβούλευση για την πρόταση τροποποίησης του άρθρου 136 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Σύμφωνα την αποστευμένη διαδικασία που προβλέπεται στο έκτο, στην έκτη παράγραφο του άρθρου 48. συνεδρίαση του 1η Φεβρουαρίου θα γίνει 1η, 1 1η Φεβρουαρίου και έκτακτη στις 17 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο. πάνω σε αυτό το θέμα. Υπενθυμίζω ότι οι συντονιστέ καθόρισαν τον υποφαινόμενο συγγητή όσον αφορά την εξέταση του σχεδίου διοργανικής συμφωνίας που αφορά το Δημόσιο Μητρό για, τις, για τη διαφάνεια όσον αφορά δηλαδή τις ομάδες συμφερόντων. Ε, αν δεν υπάρχουν παρατηρήσει όσον αφορά τι προτάσει των συντονιστών, θεωρούνται συγκεκριμένε από την Επιτροπή. Υπενθυμίζω, μεταξύ άλλων, και το εξή, ότι βάσει των συμφωνιών που έγιναν με του συντονιστέ, 27 και 28, ε, την προσωπία μα θα πάει στον Αμένα Βασίλειο. Κ. Γκαλτιόρη, Χέφνερ, Ράγκελ, Σουλ, Σταρκόφσκι και ο υποφαινόμενος θα μεταβούμε. Ο κύριος Νταφ σύμφωνα την παράδοσή μας θα συμμετάσχει ως πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρέπει να πω επικεφαλή διαπραγματευτή Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προσχώρηση τη Ευρωπαϊκή Ενώση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ελευθεριών, των θεμελιωδών ελευθεριών, ο κύριο Κρέμερ, Συνομικής ε, Υπηρεσίας θα ενημερώσει προέδρου και όλοι συγητές, συγκητές συντονιστές Επιτροπής Ελευθεριών και ΑΦΚΟ σε μια συνάντηση που θα γίνει και κλεισμένο το θηρόν στι 7 Φεβρουαρίου από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα που θα αποφασίσει όποιος αποφασίσει να συμμετάσχει μπορεί να το κάνει σαν μέλος αυτής της Επιτροπής. Φτάνει να ενημερώσει δεόντως την ε, γραμματεία. Λοιπόν, τώρα καλωσορίζω τον κύριο Γιάννη Ματώνη που είναι Υπουργό Εξωτερικών τη Δημοκρατία Ουγγαρία. Τον γνωρίσαμε μαζί με την κυρία Ένικο Γιώρη, εφυπουργό. Ήταν μέρο του Κοινοβουλίου μα παλιά και συναντήσαμε και στην Ουγγαρία όταν πήγαμε. Του συναντήσαμε και τον Προεδρεύοντα και την κυρία Υφυπουργό μετά ήρθαν εκείνοι στη διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών και μετά στο Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες τους ακούσαμε που μας μίλησαν και τους συναντήσαμε σήμερα το πρωί. Μπορούμε να ακολουθ... Όλη η Επιτροπή μπορεί να ακούσει τα προγράμματα και τις προτεραιότητες της Προεδρίας. Χαιρόμαστε που επί Ουγγρικής Προεδρίας μπορεί να υπογραφεί ο κανονισμός όσον αφορά την πρωτοβουλία των πολιτών και μπορούμε να εκφράσουμε την ευχή να προχωρήσει εντάχει κατά διάρκεια προεδρία της Ουγγαρίας η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών. Σας είπα ότι το άρθρο 136 έχει τροποποιηθεί όσο αποφασίστηκε από το Συμβούλιο και η δική μας Επιτροπή, όπως είπα και σημερομηνίας, θα προχωρήσει γρήγορα η Επιτροπή μα όσον αφορά το θέμα αυτό τη Η Εισηγητή είναι ο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη και ο Έλμαρ Μπροκ. Σήμερα το πρωί, το πρώτο σημείο τη ημερήσια διάταξη είναι οι παρεμβάσει του Προεδρεύοντο του Συμβουλίου που όπως σας είπα επανειλημμένα τον έχουμε συναντήσει και άλλες φορές και τον παρακαλούμε όμως να επαναλάβει τις προτεραιότητες το πρόγραμμα της Ουγγρικής Προεδρίας του εξαμήνου αυτού. Ευχαριστώ λοιπόν κύριε Βοντά. Έχετε το λόγο. Αγαπητά μέλη, της Επιτροπής, κύριε Πρόεδρε. Είναι μια ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμένα να έχω την ευκαιρία να σας μιλήσω και χαίρομαι για το ότι συμφωνούμε πως έχουμε μπροστά μας μια ιστορική ευκαιρία την οποία πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Δεν θα μπω τώρα στις λεπτομέρειες του προγράμματος της Προεδρίας μας. Υπάρχει χρόνο γι' αυτό. Θα ήθελα να φέρω τους βασικότερους στόχους τους οποίους έχουμε ορίσει. Όσον αφορά λοιπόν τους στόχους της Ουγγαρίας είναι σαφές πως ε, θα επιτευχθούν μόνο σε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο στενή συνεργασία Συμβουλίου Κοινοβουλίου. Ως ε, Υπουργός ε, Εξωτερικών λοιπόν και Πρόεδρευον του Συμβουλίου είναι για μένα εξαιρετικό σημαντικό να δημιουργήσουμε τις βάσεις για την ε, συνεργασία οι οποία θα πρέπει να είναι η αμοιβαία διαβούλευση και εμπιστοσύνη. Το πρόγραμμα, ξέρετε, προβλέπει πάρα πολλές διαβουλεύσεις. Έχουμε τις υπόλοιπες 26 ε, χώρες, εκπροσώπους ε, Κομισιών και Κοινοβουλίου, εκπροσώπους ε, των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, των υποψηφίων χωρών, των χωρών της Ανατολικής συνεργασίας και θέλουμε να επικεντρωθούμε λοιπόν βασικά για να επιτύχουμε το στόχο μας, το στόχο μας ο οποίος είναι μια ισχυρή Ευρώπη. Η Ουγγαρία θα ήθελε να συνεχίσει τις εργασίες που είχε ξεκινήσει το τρίο ή τρεις προηγούμενες προεδρίες ε, για να δημιουργηθούν στιβαρές θεσμικές βάσεις για την Ευρώπη. Θα θέλαμε και εμείς λοιπόν να συνεισφέρουμε στην ενίσχυση του οικονομικού συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών για τη δημιουργία μιας στέρεης βάσης για την ανάπτυξη και στόχο έχουμε να βγει η Ευρώπη ισχυρότερη στο τέλος αυτού του εξαμήνου από ό,τι είναι στην αρχή του. Μόνο μια ισχυρή Ευρώπη μπορεί να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες προκλήσεις. Η Ευρώπη μπορεί να είναι ισχυρή μόνο εάν είναι κοινά, ισχυρά τα κοινά θεσμικά μας όργανα και συνεργαστούμε για την επίτευξη αυτών των στόχων. Για τις ε, βασικές λοιπόν αποστολές ε, της Προεδρίας μας, σε αυτές δεν ανήκουν μόνο οι φάκελοι, τους οποίους ε, κληρονομήσαμε, αλλά η συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων, το πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε χωρίς μεγάλες τριβές αυτή τη συνεργασία και να καταφέρουμε να διεκπαιρεώσουμε διάφορα ζητήματα σε χρόνο ρεκόρ. Θέσαμε λοιπόν τέσσερις προτεραιότητες. Ε, προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας, καλύτερη στήριξη ε, των ε, επιχειρήσεων, κατόπιν βεβαίως ενίσχυση των κοινών πολιτικών και της ανταγωνιστικότητας, ταυτόχρονα με την διατήρηση των βασικών μας αρχών και της συνοχής. τρίτων η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πλησίασμα των πολιτών και τέταρτον η ε, υπεύθυνη συνέχιση της διαδικασίας της διεύρυνσης. Η Ουγγαρία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου σε μια αποφασιστική στιγμή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Γι' αυτό θεωρούμε πως οι προτεραιότητες που έχουμε θέσει είναι ήδη πάρα πολύ σημαντικές και ίσως σημαντικότερη προτεραιότητα είναι ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών και το πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το σχετικό νομικό πλαίσιο, αλλά πρέπει να σκεφτούμε πως τελικά υπάρχει κάτι το πολύ σημαντικότερο, το οποίο είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Γι' αυτό το σύνθημά μας είναι ισχυρή Ευρώπη με ανθρώπινη διάσταση with the human touch, όπως λέμε. Και βεβαίω ε, έχουμε κάποιες αξίες, οποίες έχουμε, τη δημογραφική αλλαγή. Και... Και ε, συνοχή, είτε μιλάμε για κοινωνικέ ομάδε, είτε για κάποιες χώρες, οι οποίες ε, θα πρέπει βεβαίως να ε, ακολουθήσουν κάποια πορεία μέχρι να φτάσουν στην ένταξη. Τώρα θα ήθελα να θέσω κάποια συνταγματικά ζητήματα. Όσον αφορά τις ε, διοργανικές σχέσεις, γνωρίζουμε πως αναδιαμόρφωσε τα πράγματα η συνθήκη της ε, Λισαβόνας σε μια άλλη επιτροπή. Εγώ ανέφερα ήδη τις ε, νομικές πτυχές, όμως θα μπορούσαμε να πούμε πως σημαντικό είναι αυτό το οποίο δεν άλλαξε, αυτό το οποίο έμεινε το ίδιο και είναι το σημαντικότερο δηλαδή μια κοινοτική μέθοδος η οποία ενισχύεται. Έχουν αλλάξει αρμοδιότητες, έχουν αλλάξει κάποιες πτυχές, αλλά η ουσία παραμένει η ίδια. Κοινοτική μέθοδος για εμένα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνεργασία θεσμικών οργάνων στο πλαίσιο που προβλέπουν οι συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, οι αλλαγές αυτές οδηγούν σε ζητήματα ερμηνείας, καμιά φορά σε διαφωνίες. Οι διαφωνίες οι οποίες βεβαίως μπορούν να αποφευχθούν και βεβαίως Το θέμα για μένα δεν είναι να υπάρχουν ερμηνεί, ε, διαφορές στις ερμηνείες και ποιος είναι ακριβώ το, το γράμμα του νόμου και των συνθήκων, αλλά το να μην εμποδιστεί η λειτουργία της Ένωσης. Και επιλέγουμε λοιπόν αυτό τον τρόπο λειτουργίας και μπορούμε να παραμερίσουμε τυχόν συγκρούσεις με υπομονή, ανεκτικότητα, κατανόηση. Οπότε θα πρέπει να παραμερίσουμε όλες τις συγκρούσεις. Σε τελική ανάλυση θα πρέπει να εμβαθυνθεί η διαδικασία της ολοκλήρωσης και να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για την Ένωση και τα κράτη της. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια να επηρεάσουν αυτά τις σχέσεις Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και να θέσουν εν κινδύνο τους κοινού μας στόχους. Θεωρώ πως οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν θα αντιληφθούν κάτι τέτοιο και δεν θα μας το συγχωρήσουν Οπότε, εάν θεωρήσουν πώς επηρεάζεται η λειτουργία της Ένωσης, το έχουμε πει, το έχουν αναφέρει πάρα πολύ, πως ε, εμείς δεν σκεφτόμαστε το κύρος όσον αφορά την άσκηση της Προεδρίας, πρέπει να λύσουμε τα διοργανικά προβλήματα, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε φιλικά το Κοινοβούλιο και ελπίζουμε από μέσα μας πώς θα μας υποστηρίξει και το Κοινοβούλιο. Και οπωσδήποτε ανάλογα θα συμπεριφερθούμε. Όταν μας χρειάζεστε θα είμαστε στη διάθεσή σας και θέλουμε να έχουμε μια επικοδομητική διαβούλευση και αυτό ισχύει σε όλα τα ζητήματα στα οποία υπάρχουν διαφωνίες. Ένα, παρά το ότι δεν είναι αυτό ίσως ο σημερινός στόχος αυτής της συνεδρίασης, σίγουρο είναι πως ε, ο... θα διατρέξουμε ένα προς ένα όλα αυτά τα ζητήματα και θα καταλήξουμε στο τέλος σε ένα συμβασμό. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής. Θα ήθελα να αφαιρθώ τώρα πιο λεπτομερώ σε τρία μόνο ζητήματα, καθώς δεν μπορώ να αφαιρθώ σε όλα. Το πρώτο θέμα στο οποίο αξίζει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο είναι οι αλλαγές της συνθήκης. Το ζήτημα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ειδικά εάν η άποψή μας είναι πως πρέπει να γίνουν αυτές οι αλλαγές με μια απλοποιημένη διαδικασία. για να μην αλλάξει ίσως η θεσμική ισορροπία. Βεβαίως κανείς δεν υπολόγιζε σε μια τέτοια αλλαγή των συνθήκων. Ετέθη ε, ενισχύ η συνθήκη της Λισαγώνας και υποθέταμε πως θα κρατήσουν λίγο χρόνο οι συνθήκες χωρίς αλλαγή, αλλά τώρα χρειαζόμαστε άλλη αλλαγή των συνθήκων. Πρέπει λοιπόν να συμφωνήσουμε πως θα πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατόν αυτές οι αλλαγές. Προσθέτω και πιθανώς το ξέρετε πως η Προεδρία εδώ πέρα παίζει αποφασιστικό ρόλο υπό την διεύθυνση της Προεδρίας θα κυλήσει όλη αυτή η διαδικασία και βεβαίως θα την υποστηρίξουμε, θα υποστηρίξουμε την αλλαγή της συνθήκης και θα προσπαθήσουμε να την περιορίσουμε στο, στη μικρότερη δυνατή έκταση. Και βεβαίως πρόκειται για ένα διακυβερνητικό μηχανισμό στον οποίο τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης θα έχουν τον πρώτο ρόλο. Η Ουγγαρία δεν είναι ακόμα μέλος της Ευρωζώνης και δεν μπορούμε να πούμε πότε θα γίνουμε, αλλά σίγουρο είναι πως έχουμε δώσει το μήνυμα στα υπόλοιπα ε, κράτη-μέλη πως οπωσδήποτε θα συμπεριληφθούν και μη κράτη-μέλη της Ευρωζώνης στην διαδικασία αυτή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως υπάρχει μια σχέση μεταξύ αλλαγής της συνθήκης και άλλων θεμάτων. Και εδώ, κατά κύριο λόγο, μιλάμε για την δημιουργία των κανόνων, για την φορολογία των επιχειρήσεων και βεβαίως πρέπει να δούμε πως ε, η Ουγγαρία θα πρέπει να δει αυτά τα δύο θέματα με έναν πιο υγιή τρόπο. Γιατί ξέρετε αυτές οι συνδέσεις καμιά φορά οδηγούν σε νομικούς κινδύνους. Τώρα κάποια λόγια για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών. Η σημασία αυτού του θέματος πηγαίνει πολύ πιο πέρα από αυτά τα οποία είχαμε σκεφτεί αρχικά όταν ε, εγκρίθηκε στην συνθήκη της Λισαβόνος η πρωτοβουλία αυτή. Προσπαθούμε λοιπόν να μειώσουμε το δημοκρατικό έλλειμμα για το οποίο μιλούσαμε εδώ και δεκαετίες. Υπάρχει λοιπόν μια ενότητα και εκτιμούμε πάρα πολύ τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου που οδήγησε σε αυτή την ενότητα και νομίζω πως είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα παραμέρισης των διαφορών μας και για το πώς μπορούν να λυθούν ή διαφορές λογικά. Αυτό συνέβη και είναι κάτι το οποίο χαιρετίζουμε και βεβαίως η διαφορές λογικά. Αυτό συνέβη και είναι κάτι το οποίο χαιρετίζουμε και βεβαίως αποστολή μας τώρα είναι να εφαρμοστεί και στην πράξη το συντομότερο δυνατόν η πρωτοβουλία των πολιτών. Ελπίζουμε στις 14 Φεβρουαρίου το Συμβούλιο να εγκρίνει την πρόταση και η Ολομέλεια μετά του Κοινοβουλίου να εγκρίνει αυτές τις ε, αλλαγές. Αυτό σημαίνει πως ήδη θα τεθεί ενισχύει ο κανονισμός επί Ουγγρικής Προεδρίας και θα μπορεί να ξεκινήσει η περίοδος του ενός έτους και να έχουμε αυτό το μέσο άμεσης δημοκρατίας στην πράξη. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΕΣΔΑ. Αλλά βεβαίω η συνθήκη δεν ήταν το κατάλληλο μέσο για να λυθούν όλα τα λεπτομερή δήματα που ανέκυψαν π.χ. τι θα γίνει με τους ε, πιθανούς ε, αντιδίκους σε μία υπόθεση, ποιος θα εκπροσωπεί την κοινότητα, αν θα είναι η Κομισιόν, ή όχι. Εμείς λοιπόν θα, θα ρίνουμε τα κράτη με να υποστηρίξουν αυτές τις διαπραγματεύσεις και είμαι πεπισμένος πως όλα τα νομικά προβλήματα θα μπορέσουν να ξεκαθαρίσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ουσιαστική σημασία εδώ πέρα έχει το να εκμεταλλευτούμε το ότι προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης εξακολουθούμε να Θεωρούμε, όπως και πριν, πως όλα τα επίμαχα μπορούν να λυθούν μέσω του διαλόγου. Και αυτό ισχύει για τις ε, διαπραγματεύσεις μέσω το, ε, τις διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τις προοπτικές. Είχαν ήδη ξεκινήσει και ελπίζουμε πως σύντομα θα έχουμε συγκεκριμένες ε, προτάσεις. Επιτάπητος θα ασχοληθούμε λοιπόν και με ζητήματα τα οποία αφορούν τις ε, διαπραγματεύσεις. Πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε σε μία λύση αποδεκτή από όλα τα μέρη και γνωρίζουμε πως πρέπει να ασχοληθούμε και με το θέμα της πρόσβασης στα ε, έγγραφα. Όπως σας είπα, όλα αυτά θα λυθούν μέσω διαβουλεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε σίγουροι λοιπόν πως θα έχουμε επιτυχία γιατί είναι προς το κοινό μας συμφέρον και αφορά βεβαίως και την επιτυχή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα αυτά τα ζητήματα. Η Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων έχει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε ολόκληρη την περίοδο της Προεδρίας μας. Γι' αυτό σας παρακαλώ εσάς, τα μέλη της Επιτροπής, να μας στήριξετε σε αυτό. Και ζητώ ιδιαίτερα τη δική σας στήριξη, γιατί η επιτυχία της ε, Ουγγρικής Προεδρίας θα ε, υπάρξει μόνο σε συνεργασία με την Επιτροπή σας. Είμαι λοιπόν έτοιμος για αυτή την συνεργασία και αυτή την καλή θέληση εραμένω και από σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Βόντα. Ευχαριστώ κύριε Πρεδρεύοντα. Οι συνάδελφοι θα μιλήσουν για να ζητήσουν κάποιες διευκρινήσεις ή για να υπογραμμίσουν κάποιες πτυχές. Πρώτα απ' όλα όμως θα ήθελα να ζητήσω από την Υφυπουργό, την κυρία Ινίκο αν θέλει να προσθέσει κάτι. Δεν επιθυμείτε να μιλήσετε. Καλώς μπορείτε να μιλήσετε κατά τη διάρκεια της συζητήσεως. Καταρχάς, έχω μία ερώτηση, κύριε Προεδρεύοντα. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός, ο κ. Όρμπαν, αναφέρθηκε και στη διεύρυνση και στην προσχώρηση της ε, Κροατίας σαν προοπτική να γίνει σύντομα η προσχώρηση της Κροατίας στην Ένωση. Ή δυνατόν θα μπορούσατε να μας πείτε πότε κάποιο χρονοδιάγραμμα ώστε αυτή η Επιτροπή να λάβει τα δέοντα μέτρα. και ε, να έχουν κάποιο προσανατολισμό και ενόψη και των προσεχών ευρωεκλογών του 2014, συνάδελφοι. Ε, Σάιγερ, ο κύριος Σάιγερ έχει το λόγο πρώτος ο συναδέλφος. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς ως Ούγγροι χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την ανάληψη της Προεδρίας γιατί εάν είχε επιτύχει η επανάσταση του 56 θα ε, ήμασταν στα ιδρυτικά μέλη της Ένωσης, αλλά ξέρετε και εσείς πως η ιστορία κύλησε διαφορετικά. Βεβαίως, για χώρες που έχουν ασκήσει πολλές φορές την Προεδρία δεν είναι και τίποτα το σπουδαίο, αλλά εμείς ως Ούγγροι το βλέπουμε ακόμα ως κάτι το μεγάλο και σπουδαίο. Σας καλωσορίζω λοιπόν. Είστε ένας από τους λίγους Ευρωπαίους ε, πολιτικούς ε, που ε, επιθυμούν να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντα της χώρας τους βεβαίως αλλά και τα συμφέροντα της Ευρώπης. Σύντομα λοιπόν για το βιογραφικό. Την ε, ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με συγχωρείτε τώρα που αναφέρομαι προσωπικά στον κύριο Υπουργό, αλλά όλα αυτά σχετίζονται άμεσα με την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν λοιπόν παρόν σε όλα τα σημαντικά γεγονότα 1990-94 όταν καταθέσαμε την αίτηση ένταξης στην διάρκεια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων ήταν διαπραγματευτής ε, και υπουργός την εποχή εκείνη. Επίσης στην συνέλευση, την συντακτική είχε απευθυνθεί στην ε, Ολομέλεια όχι μόνο ως ε, υπουργός αλλά και ως εμπειρογνώμονας. Βοήθησε πάρα πολύ στις εργασίες. Και τώρα, όπως ξέρετε, ε, ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου. Και το ότι είμαστε εδώ πέρα, όπως είπα, είναι για εμάς μια μεγάλη ικανοποίηση. Αξιότιμοι συνάδελφοι, τώρα σε σχέση με την αλλαγή της συνθήκης θα ήθελα να πω πως ο κύριος Υπουργός μιλά ενώπιον συναδέλφων και έχουμε μπροστά μας ε, να αντιμετωπίσουμε ζητήματα, πάρα πολλά ζητήματα, πάρα πολλά σημεία στα οποία πρέπει να αλλάξει η συνθήκη. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως πως θα διατρέξουμε έναν κατάλογο ή μια ολόκληρη λίστα, αλλά θα πρέπει να περιοριστούμε σε λίγα μόνο σημεία. Επίσης θεωρώ πως όταν επιτέλους ολοκληρωθεί αυτή η συνθήκη θα πρέπει να την αφήσουμε λίγο στην ησυχία τους. Υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν μπορούν να αλλάξουν το σύνταγμά τους τόσο γρήγορα. Βεβαίως, εάν είναι αναγκαίο για να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή συνεργασία, θα πρέπει να μπορεί να επαναληφθεί η διαδικασία. Ακούσαμε πως η Προεδρία θέλει να είναι φιλική προς το Κοινοβούλιο. Ε, δεν είναι ωραίο να έχουμε τόσο πολλές διοργανικές συγκρούσεις. Καλό είναι να έχουμε μια συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και βεβαίως για τους πολίτες σημασία έχει να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, δεν έχει σημασία, τους ενδιαφέρει η διαδικασία. Όσον αφορά δε την επιτροπολογία, εμένα με ενδιαφέρε πάντα και βέβαια και τους ε, διάφορους πίνακες ε, που αναφέρθηκαν από τον κύριο Υπουργό της πίνακης αντιστοιχίες αλλά μπορούμε να αναφέρουμε και θετικά παραδείγματα. Π.χ. ο κύριος Όρμπαν την προηγούμενη εβδομάδα είπε για το έλλειμμα του προπολογισμού πώς θα δώσει το καλό παράδειγμα. Η Ουγγαρία υπάρχει ήδη μια συζήτηση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για αυτό το θέμα και νομίζω πως εάν πάνε καλά αυτές οι συνομιλίες θα δημιουργήσουμε μια σχολή. Αυτό βεβαίω δεν είναι αυτός ο σκοπός, πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου τα συμφέροντα των πολιτών. Ακούσαμε επίσης πώς μπορούμε να απευθύνουμε ερωτήματα στον κύριο Υπουργό και το ερώτημά μου αφορά ακριβώς αυτούς τους πίνακες αντιστοιχίας και σας εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας. Σας ευχαριστώ κύριε Σάγερ. Και εγώ, όπως και άλλες φορές το έκανα, θα ήθελα να εκφράσω τη συγκίνησή μου έναντι της Ουγγρικής Προεδρίας, που με φέρνει πίσω στη νεότητά μου. Η επανάσταση του 56 φαινόταν η μάχη του Δαβίδ κατά του Γολιάθ και εμεί καθόμασταν και βλέπαμε, μην μπορώντα να κάνουμε κάτι για προφανεί λόγου, για την παγκόσμια ειρήνη. Και είναι ε, συγκλονιστικό που σήμερα η Ουγγαρία ηγείται της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και εγώ υπογραμμίζω λοιπόν αυτό που είπατε κι εσείς. Γνωρίζω το ότι μετά στις 10.30 πρέπει να περάσουμε στην ακρόαση των εμπειρογνωμόνων και πολιτικών προσωπικότητων όσον αφορά το καθεστώς, τη χρηματοδότηση των ε, πολιτικών κομμάτων. Θα ήθελα να ζητήσω από τους παρεμβαίνοντες, που είναι πολλοί, να συγκρατηθούν στα τέσσερα 4 λεπτά για κάθε παρέμβαση. Ο κύριος Ντάφ έχει ζητήσει το λόγο. Um, Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά και αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά για την ευκαιρία που έχουμε να υποδεχθούμε τον Ούγγρο Πρόεδρε, τον Ούγγρο Υπουργό. Εμείς, ε, οι πρεσβύτεροι δηλαδή της συντακτικής συνέλευσης, έχουμε μία λέσχη μεταξύ μας και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως όταν ε, ασχολούμαστε με τέτοια συνταγματικά ζητήματα. Δύο σχόλια. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την οικονομική διακυβέρνηση και το προσωπικό. Όπως ξέρετε, υπευλήθη έτοιμα για έγκριση μιας ε, έκτακτης καταξαίρεση διαδικασίας για τις ε, προτινόμενες αλλαγές στη συνθήκη της Λισαβόνας. Εγώ προσωπικά αλλά και η ομάδα μου δεν πιστεύουμε ότι οι προτινόμενες αλλαγές αρκούν μακροπρόθεσμα για την ε, εξασφάλιση μιας αξιόπιστης ε, οικονομικής κυβέρνησης. Αυτό το αντιλαμβάνονται και οι αγορές. Και όλο και περισσότερο αρχίζουν και το αντιλαμβάνονται και οι πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξετάσει αυτό το θέμα και μάλιστα ο εισηγητή μας για το ζήτημα αυτό θα είναι ο κ. Γουαλτιέρη, θα το σχολιάσει φαντάζομαι. Κατά πάσα πιθανότητα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προσεγγίσει αυτό το θέμα ως πρώτο βήμα μόνο, ως το σημείο αφετηρίας και αναμένουμε μία ολόκληρη σειρά διαδοχικών αλλαγών που θα προταθούν μέσο και μάκρο πρόθεσμα. Και ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ταχθεί υπέρ ενό τέτοιου αποτυπώματο ό,τι αφορά τα κριτήρια σύγκλησης. Ε, αυτή η πρόταση πιστεύω ότι μπορεί να μας μεταφέρει από το σημερινό σημείο, από τη σημερινή κατάσταση σε μια πιο γνήσια οικονομική κυβέρνηση με χαρακτηριστικά και Δημοσιονομικής Ένωσης. Και ελπίζω ότι η Ουγγρική Προεδρία θα ενθαρρύνει και θα προωθήσει μια τέτοια συζήτηση. Στο Συμβούλιο βέβαια κάποιοι ομόλογοι σας θα αντιταχθούν στεναρά α, ακόμη και ως προς τη διοργάνωση μιας τέτοιας συζήτησης για τα πιο θεμελιώδη ζητήματα της οικονομικής διακυβέρνησης. Ευελπιστώ πάντως ότι η Ουγγρική Προεδρία θα μπορέσει να αξιοποιήσει και την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να την εκμεταλλευτεί κατά κάποιο τρόπο για να ενισχύσει το επιχείρημα της δημοκρατικής προσέγγισης αυτού του προβλήματος, της ενίσχυσης της σταθερότητας των οικονομικών μας και του συνδυασμού τους με την προσπάθεια οικονομικής ανάκαμψης. Σε ό,τι αφορά την ε, δημοσιονομική μεταρρύθμιση, τη μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού και την κατάρτιση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, καθώς και την αναθεώρηση του συστήματος ιδίων πόρων, κατά τη γνώμη μου είναι κέρια σημασία να συμμετέχει πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη συζήτηση αυτή. Γιατί αν αποκλειστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή παραμεληθεί, παραγωνιστεί. Πιστεύω ότι η έκβαση των συζητήσεων, που ούτως ή άλλως θα είναι ακαθόδης και αρκετά χρονοβόρες, μπορεί να αμφισβητηθεί. Δεν νοείται μία αίσια έκβαση αυτών των διαπραγματεύσεων με αποκλεισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ε, πλήρη και αμέριστη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή. Βλέπω να δυσανασχετεί ο Πρόεδρος με την παράταση του χρόνου αγόρευσης. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να ολοκληρώσω. Σε ό,τι αφορά την εκλογική μεταρρύθμιση για τις ευρωεκλογέ. Και για αυτό το θέμα εκδήλωσε ενδιαφέρον η Ουγγρική Προεδρία και ελπίζω ότι κατά την Άνοιξη θα ψηφίσουμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα ευρύτατο πακέτο, μια δέσμη μέτρων για την ε, μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας και για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή την πρόταση θα την υποβάλουμε και στον πρόεδρο Βαν Ρομπό, γιατί απαιτούνται κάποιες μικροαλλαγές στη συνθήκη γι' αυτό. Πάντως θα πρέπει και το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ε, να εξετάσει αυτή την πρόταση και να λάβει θέση. Πολύ θα με ενδιαφέρει λοιπόν η εθερμό αντίδραση του Υπουργού Ματώνη για τις προτάσεις που αυτή τη στιγμή εξετάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς την εκλογική μεταρρύθμιση. Ευχαριστώ κύριε Ντάφ. Πράγματι άρχισα να δισταρισχετώ, να ανησυχώ, αλλά όμως θα κλέψω λίγα λεπτά για να ευχηθώ, γιατί χτες ήταν τα γενέθλιά σας. Λοιπόν, σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και θα να σας πω τις σκέψεις σας όσον αφορά τις ε, τροποποίησεις της συνθήκης, της ενώσεως. Είναι σωστές, οι σκέψεις σας είναι σωστή και προβλέπεται από τη συνθήκη. Ε, τρεις φορές το προήμιο στο άρθρο 1 επίσης αναφέρεται σαν βήμα και σαν διαδικασία. Λοιπόν, θα πρέπει συνεχώς να γίνονται οι προσαρμογές, χωρίς να ανησυχούμε και να τρομάζουμε. Ο κ. Μέντες Δεβίγου έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ευκαιρία συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων με τον Υπουργό Μαρτώνη. Θα είμαι λακωνικότατος ε, για να δημιουργήσω και κάποιο προηγούμενο, γιατί αλλιώ ε, θα εξαντλήσουμε το χρόνο και θα προλάβουμε να συζητήσουμε. Αυτό το θέμα το 136 είναι η δεύτερη αλλαγή της συνθήκης της Λισαβόνας. Αλλά τι έγινε με την πρώτη αλλαγή σε ό,τι αφορά την επικύρωση του πρωτοκόλλου 36. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Ουγγρική Προεδρία να ε, παροτρύνει τους πιο οκνηρούς αυτή τη διαδικασία επικύρωσης ε, να σπεύσουν και να ολοκληρώσουν την επικύρωση του πρωτοκόλλου 36. Ό,τι αφορά την τροποποίηση του 136, πιστεύετε ότι στην έκθεση Μπροκ και Γουαλτιέρη, καλό θα ήταν να έχουμε μια πλήρη επισκόπηση των φιλοδοξιών μας για την οικονομική διακυβέρνηση, μια και ο, ο μόνιμος μηχανισμός σταθερότητας είναι ένα και μόνο τμήμα, σημαντικό μεν, αλλά ένα και μόνο τμήμα του συνολικού οικοδομήματος αυτής της οικονομικής διακυβέρνησης. Σας ευχαριστώ για την λακωνικότητά σας. Γκουερέρο. Σας Γκουερέρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς εγώ δεν θα καταφέρω να είμαι τόσο λακωνικός σαν τον κύριο Βίγκο. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Υπουργό Μαρτών, να τον ευχαριστήσω για την παρουσία του εδώ και να τον συγχαρώ για την πρώτη φορά που η Ουγγρική Προεδρία θα σκίσει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί η Ουγγαρία ήταν μια χώρα που έχασε την δημοκρατία αλλά κατάφερε να την ε, ανακτήσει και φαντάζομαι την υπερηφάνεια που θα αισθάνεστε για κάτι τέτοιο. Και εγώ θυμάμαι το ρόλο μου την πρώτη φορά που άσκησε η Ισπανία την ε, Προεδρία και τότε ήμουν επικεφαλής του γραφείου του κ. Σολάνα και πραγματικά η εμπειρία μας ε, θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη μας. Γι' αυτό σας συγχαίρω θερμά για την παρθενική σας Προεδρία. Εκ μέρου ε, των Σοσιαλιστών και των Δημοκρατών θα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη υποστήριξή μου προς τους στόχους ε, και τις προτεραιότητες της Ουγγρικής Προεδρίας, γιατί η επιτυχία της ε, Ουγγρικής Προεδρίας θα είναι επιτυχία ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει θετική αντανάκλαση σε όλες τις χώρες μέλη. Θα ήθελα να επισημάνω ορισμένα από τα θέματα που αναφέρομαι. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την προσπάθεια προώθησης ε, της ε, έμπρακτης εφαρμογής της πρωτοβουλίας των πολιτών, γιατί δεν θα πρέπει μόνο να εφαρμόσουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά να ικανοποιήσουμε και την επιθυμία των Ευρωπαίων πολιτών για ενεργό συμμετοχή τους στον πολιτικό βίο της Ένωσης. Γιατί πρόκειται για κάτι που έχει Γάλλο πατέρα και Ουγγαρέζα μητέρα και κατά κάποιο τρόπο η Ουγγαρία έχει δεσμευθεί υπέρ της ανάπτυξης αυτής της πρωτοβουλίας των πολιτών. Σε ό,τι αφορά την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την οποία είμαι συγγετής, μέσα σε δύο εβδομάδες θα έχουμε και πάλι τον διαπραγματευτή εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη συνεδρίασή μας για να μας ενημερώσει για τις λεπτομέρειες των διαπραγματεύσεων το μόνο που μπορώ να ζητήσω είναι ότι αν έρθουν σε αίσιο πέραση διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Ουγγρική Προεδρία καλό θα ήταν να προωθήσει την έγκρισή του στο Συμβούλιο και την μεταγενέστερη κύρωση της ε, συμφωνίας αυτής από τα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές προοπτικές, Ξέρω ότι ακόμη δεν τις έχετε εντάξει στο πρόγραμμά σας, αλλά στα πλαίσια των τριών διαδοχικών προεδριών και των συναντήσεών τους, καλό θα είναι να αρχίσετε να εξετάζετε και το σημείο αυτό. Και θα ήθελα να αφιερώσω και ένα λεπτό σε κάτι που μου είναι ιδιαίτερα προσφυλές, γιατί ως πρώην μέλος της Επιτροπής Στεγματικών Υποθέσεων και στην Ισπανία, Είχαμε συνάντηση παρουσία για τον κύριο Σόφλιν και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συζήτηση για τα θέματα αυτά και ξέρουμε ότι και στην Ουγγαρία έχει ξεκινήσει μια ε, διαδικασία συνταγματική αναθεώρηση γιατί η Ουγγαρία είναι η μοναδική χώρα που δεν έχει αναθεωρήσει το σύνταγμά τη από την απολυταρχική περίοδο τη πολιτική τη ζωή. και έχετε τώρα την ευκαιρία να μετατρέψετε το νέο σα σύνταγμα σε ένα δημοκρατικό ε, σύνταγμα κατοχύρωση με μελιωδών δικαιωμάτων έναν του προηγούμενου συντάγματος. Και μάλιστα η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης στηρίζεται στην ε, υποστήριξη των πολιτών σας, όπως προέκυψε από την εκλογική διαδικασία. Εγώ δεν θα κάνω αξιολογικές κρίσεις για την αναθεώρηση αυτή. Έχετε διπλή ιδιότητα πάντως αυτή τη στιγμή, την ιδιότητα του Προεδρεύοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την ιδιότητα του ε, Ουγγρου Υπουργού. Θα ήθελα να ενοποιήσετε αυτές τι δύο ιδιότητε αν γίνεται, και οι αρχές που θα προασπίσετε εδώ να είναι οι ίδιες με αυτές που θα προτάξετε και θα υπερασπίσετε και στη χώρα σας. Λοιπόν, διαβούλευση, αμοιβαία, ε, αμοιβαία συνεργασία, ανοχή, ενσυναίσθηση, κατανόηση, αμοιβαία διάλογο. Νομίζω ότι αυτό είναι ο δρόμο για να καταλήξουμε σε πολιτική συνένεση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Δεν πρόκειται εγώ να επισέλθω στα εσωτερικά της πολιτικής ε, ζωής της Ουγγαρίας. Απλώς ήθελα να επισημάνω αυτές τις ε, αρχές και τις αξίες που αισθενιζόμαστε όλοι, φαντάζομαι και εσείς, και γύρω από αυτές τις αρχές θα πρέπει να οργανώσουμε τον πολιτικό μας βίο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Γκορέρο. Η κυρία Λεγκρίπ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω κύριε Υπουργέ, κυρία Υφυπουργέ για την παρουσία σας εδώ ανάμεσά μας σήμερα το πρωί και τα άκρως ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπατε, τα ισχυρά, τις δυνατές εκφράσεις που χρησιμοποίησατε, αυτά που μας είπατε, την ευκαιρία της πρώτης αναλήψεως των καθηκόντων σας στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενώσης. μεγάλη τιμή για μια χώρα αυτό. Και χαίρομαι που αυτό συνέβη στην Ουγγαρία. Και πιστέψτε με ότι καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσης ε, δεν είναι που δεν δεν δέχεται χωρίς ε, να αισθάνεται περήφανη το να είναι στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι μεγάλη ευθύνη αυτή, πολύ σοβαρό το καθήκον. Θα έχετε μεγάλη υποστήριξη ο φάσης βασικού άξονα τη Προεδρία σα τη Ουγγρική και σα έχουμε εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη είναι βασικό χαρακτηριστικό του ευρωπαϊκού προγράμματο, εμπιστοσύνη μεταξύ κρατών μελών, μεταξύ λαών και βεβαίω εμπιστευόμεθα την Ουγγρική Προεδρία. Συμμεριζόμαστε, για μία ακόμη φορά το λέω αυτό, ε, Τι μεγάλε προτεραιότητε. Θα είμαι πολύ γρήγορη για τα δύο θέματα που θέλω να αναφέρω, που ήδη αναφέρθηκαν από κάποιου κάποιους Κυρίω κυρίως το θέμα τη διευρύνσεω, που αναφέρθηκε ήδη από τον Πρόεδρο Κασίνη. Θα ήθελα να εκφράσω κάποιες παρατηρήσεις συνετέ, θα έλεγα, προσεκτικέ όσον αφορά την διεύρυνση, τη δικασία τη διεύρυνση. Θα σα ρωτήσω ποιο ήταν το χρονοδιάγραμμα. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Σα κρύβω ότι οι κοινέ γνώμες σε κάποια κράτη-μέλη όσον αφορά τη διεύρυνση είναι περισσότερο από διστακτικές. Υπάρχει σκεπτικισμός στην κοινή γνώμη κατά πόσο είναι επίγονα είναι κάτι και κατά πόσο συμφέρον να γίνουν οι επόμενες διευρύνσεις. Αυτό είναι το πρώτο που σας ρωτώ. Δεύτερο θέμα που αναφέρθηκε από τον συνάδελφο Ερέρο ήταν της θεματικής αναθεωρήσεως του συντάγματος της Ε, είχα πάει με την αντιπροσωπεία εγώ στη Βουδαπέστη, έγινε ανταλλαγή απόψεων επ' αυτού του θέματο με πολλού συνομιλητέ. Κάποιο χρονοδιάγραμμα έχετε να μα δώσετε όσον αφορά την ανεθόρυση Συντάγματο Ουγγαρία η Ουγγρική Προεδρία, μακάρι να είναι μια χρήσιμη Προεδρία, δεν μπορούμε να χρονοτριβούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω προκλήσεων κατεπηγόντων προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Θα πρέπει να είναι χρήσιμη για την Ένωση λοιπόν η Ουγγρική Προεδρία και δεν το αφισβητούμε ότι θα είναι με τη συνδρομή όλων. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. κυρία Sok szeretettel köszöntöm. Valóban nekünk lehetőségünk volt érzékelni azt, hogy ez egy... Ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλωσορίσω και εγώ θερμότατα τον Υπουργό Μαρτώνη και ήδη διστανόμαστε τη φιλική στάση της Ουγγρικής κυβέρνησης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και της Ουγγρικής Προεδρίας. Γιατί η σημερινή ομιλία του Υπουργού ήταν ένα πολύ σημαντικό μήνυμα προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί όλα τα θεσμικά όργανα έχουν τη θέση τους σε αυτή τη διαδικασία και έχουν αντίστοιχο έργο να επιτελέσουν. Η πρωτοβουλία των πολιτών είναι προτεραιότητα της Ουγγρικής Προεδρίας, όπως ακούσαμε, και είναι ένα θέμα που το επισήμανε και οι συνάδελφοι. Στη δική μας επιτροπή και ο κύριος Λαμασούρ και εγώ είχαμε αναλάβει αυτή την έκθεση για την πρωτοβουλία των πολιτών. και μάλιστα η Ισπανική Προεδρία έκανε ένα προπαρασκευαστικό έργο για την έκθεση αυτή που ήταν πολύ αξιόλογο και χάρη σε αυτή την προεργασία είχαμε το πρώτο έγγραφο στις 22 Ιουλίου κατόπιν ανέλαβε τη σκητάλη η Βελική Προεδρία και συνέχισε με την ίδια θέρμη ε, την πρόθεση αυτού του ζητήματος και η Ουγγρική Προεδρία συνεργάστηκε στα πλαίσια του τρίου των Προεδριών. Είχαμε από στις 22 Ιανουαρίου μια νέα πρόοδο και μάλιστα το γεγονός ότι η πρωτοβουλία των πολιτών απέκτησε σάρκα και ωστά χάρη στην υποστήριξη των πολιτικών κομμάτων είναι πολύ θετικό η διαδικασία είναι χρονοβόρα. Και τελικά χρειάστηκε να περιμένουμε 20 ολόκληρους μήνες για την ε, εφαρμογή της πρωτοβουλίας αυτής. Θα πρέπει τώρα αυτό το εργαλείο, η πρωτοβουλία των πολιτών, να στεφθεί με επιτυχία και να χρησιμοποιηθεί ευρέως. Η Ουγγρική Προεδρία πάντως φαίνεται ότι είναι πολύ δυναμική Και... Και βεβαίως ε, ξέρετε πως ε, το Μάιο είχαμε, θα, είχαμε ταξιδέψει και στις περιφέρειες και ξέρουμε πως ε, κατανοεί αυτά τα ζητήματα. Ο κ. Υπουργό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κάτι το νέο και βεβαίως η διαρκής συνεργασία υποστηρίχθηκε και από τους σοσιαλιστές. Ε, και έχουμε το... νομοθετικό πρόγραμμα το οποίο αναπτύχθηκε και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δύο ακόμα παρατηρήσεις. Είναι σαφές πως η Ουγγαρία αναλαμβάνει την Προεδρία σε μια σημαντική, για να μπω, ιστορική, στιγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μια πρώτη αξιολόγηση της χάρτας θεμελιωδών δικαιωμάτων και θα ήθελα να μάθω πώς βλέπει αυτή την αξιολόγηση η Ουγγρική Προεδρία και ένα θεωρητικό ερώτημα με το οποίο θα ήθελα να κλείσω. Ναι τις υποψήφιες χώρες. Υπάρχουν κάποια κριτήρια που πρέπει να εκπληρωθούν και θα ήθελα να ακούσω εάν σκέφτεστε να δούμε το νομικό πλαίσιο όσον αφορά την διεύρυνση προς Ανατολάς. Βεβαίως στην Κροατία μια τέτοια ένταξη θα θεωρηθεί επιτυχία εάν ολοκληρωθεί η Επικουρικής Προεδρίας θα είναι κάτι το πολύ καλό και βεβαίως ε, θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί σωστά η ένταξη της Κροατίας. Έχουμε συνεργαστεί επί μακρόν ε, και μπορώ άρα να βεβαιώσω πως είστε ε, Ευρωπαίος πραγματικά και Κύριε Υπουργέ, στην παρουσίασή σας Λοιπόν, έχουμε, βλέπετε, μία αλλαγή των ισορροπιών της εξουσίας, γιατί ε, με την πρωτοβουλία των πολιτών οι πολίτες έχουν εξίσου μεγάλη εξουσία με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.

Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να δώσω τις καλύτερες ευχές μου στον, ε, στον Υπουργό της Ουγγαρίας. Θα ήθελα να μπω στο θέμα της μεταρρύθμισης της συνθήκης κατευθείαν. Ο κύριος Υπουργός αναφέρθηκε στην δυνατότητα προσφέρεται μέσω της απλουστευμένης διαδικασίας και άλλοι συνάδελφοι τοποθετήθηκαν, ξέφρασαν κάποιες απόψεις. Θα έχουμε τη δυνατότητα να εμβαθύνουμε στη συζήτησή μας, σίγουρο είναι αυτό. Εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις. Με το Συμβούλιο θα έχουμε αποφάσεις, είναι ο συνομιλητής, ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μάλλον περισσότερο συνομιλητής μας για αυτό το θέμα από ότι το Συμβούλιο αλλά καλό θα ήταν να το συζητήσουμε και τώρα και με την Προεδρία την Ουγγρική. Έχω τα ερωτήματα. Σχετικά με την ε, ε, διαδικασία που θα ακολουθηθεί και ποια μεταρρύθμιση τίθεται ο στόχος. Πιστεύουμε ότι η νομισματική πολιτική των χωρών της Ευρωζώνης είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και μια ενδεχόμενη αποκέντρωση της δυνατότητας με κάποια κράτη-μέλη ομάδα 100 μελών να μπορούν να κινηθούν εκτός αποκλειστικής ε, αρμοδιότητας ε, χωρίς να απαιτείται απαραίτητα μια μεταρρύθμιση των συνθήκων. Η διαδικασία η ευέλικτη που, που προβλέπεται από τη συνθήκη δείχνει κάποιο δρόμο για ενδεχόμενη μεταρρύθμιση της συνθήκης που θεωρείται αναγκαία και πολιτική χρειά τώρα στο ερώτημά μου. Τι προβλέπετε να κάνετε σε περίπτωση προβλήματος όσον αφορά κύρωσης από τα 27 Εθνικά Κοινοβούλιο. Ο κύριος Μέντες Δεβίγο το ανέφερε τι γίνεται με την ε, κύρωση της άλλης μεταρρύθμισης. Είναι ένα πρόβλημα που ενδιαφέρει κυρίως και κάποιους ενδεχόμενους και μελλοντικούς συναδέλφους. Τι θα συνέβαινε. Η Ευρώπη θα μπορέσει να έχει κάποιο μηχανισμό διαφύλαξης, αν θέλετε, που θα προστατεύει το ενίο νόμισμα. Όσον αφορά το περιεχόμενο της μεταρρύθμισης που προτείνεται, ο συνάδελφος Νταφ μίλησε για ανεπαρκές βήμα. Σκέφτομενος το προτινόμενο κείμενο διερωτώμε αν είναι όχι ανεπαρκές βήμα, αλλά βήμα επαναχώρησης, οπισθοχώρησης ότι δεν θα μας επιτρέψει να έχουμε μια πιο σωστή δομή της διακυβέρνησης. Ο, όπως έχει πρόταση του μηχανισμού σταθερότητας που έχει διακυβερνητική χρειά, που δείχνει ότι ενώ το σημερινό, το προσωρινό που χρησιμοποιείται μηχανισμός της Ένωσης, διότι άπτεται και του προπολογισμού, δεν έχουμε τη δυνατότητα στο μέλλον να έχουμε σαν πολιτική της Ένωσης μηχανισμό σταθερότητας. Λέμε ότι από τούτο και στο εξή ένας μηχανισμός σταθερότητας θα μπορεί να εφαρμόζεται μόνο από μια ομάδα χωρών εκτός της δομής της Ενώσεως χωρίς να υπάρχει ρόλος για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα θεσμικά όργανα της Ενώσεως, συμπεριλαμβανομένου και του Κοινοβουλίου. Δηλαδή, αντί να δημιουργούμε μια δυνατότητα, δημιουργούμε ένα δεσμό. Είναι αρνητική η προσέγγιση όσον αφορά τη δυνατότητα να δράσουμε στο μέλλον. Λέμε ότι δεν θα μπορέσουμε πλέον ποτέ να δημιουργήσουμε μηχανισμό τη Ένωση για σταθερότητα τη Ευρώπη. Θα πρέπει να το κάνουμε σαν μηχανισμό μια ομάδα κρατών μελών εκτό τη Ενώσεω. Είναι μια σοβαρότατη ευθύνη αυτή το να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο. Και αμφισβητώ ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε δρόμο που μας οδηγεί προς τα πίσω να μας πει λοιπόν ο κύριος Υπουργό κατά πόσο υπάρχει προβληματισμός επί του θέματος και ποια είναι η άποψή του όσον αφορά συγκεκριμένο ζήτημα. Ευχαριστώ κύριε Γκουαλτιέρη. Ο κύριος Βερκόσκη, ο αντιπρόεδρος, συνάδελφος, έχει το λόγο. Κύριε Υπουργέ, προσωπικό σχόλιο, την εποχή την κομμουνιστική, μας δίδασκαν διαφορετικές εκδοχές της ιστορίας από ό,τι μας μάθανε η πραγματικότητα. Μου μάθανε ιστορία ο πατέρα μου στο σπίτι και όταν σχολίαζε το 15ο αιώνα, όταν η Ουγγαρία και η Πολωνία ε, συνδεόταν με δυναστικούς δεσμού. Ε, αναφερόταν στο πώ επηρεάζουμε τα χτενόμενα τη Ευρώπη. και έλεγε η ιστορία δεν σου δίνει ποτέ δεύτερη ευκαιρία και αυτό μου το έλεγε εδώ και 20 χρόνια. Συγκινήθηκα όταν αναλαμβάνατε την Προεδρία διότι νομίζω η ιστορία μα δίνει μια δεύτερη ευκαιρία να επηρεάσουμε τη διαδρομή τη Ευρώπη. και γι' αυτό σας εύχομαι ένθερμα τεράστια επιτυχία στην Προεδρία σα. Έχω δύο ερωτήσει. Η μία είναι αρκετά αφελή, διότι είστε διπλωμάτη, οπότε πιθανότατα θα πρέπει να πείτε ότι η συνεργασία είναι υπέροχη και δεν υπάρχουν προβλήματα. Σας ρωτήσω παρόλα αυτά τι γίνεται με τη συνεργασία με την, καθ... με την κυρία Άστον εν την προετοιμασία της Προεδρίας κυρίως όσον αφορά την κατανομή των αρμοδιοτήτων, το μοίρασμα της δουλειάς και τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και άλλα τεινά. Και όσον αφορά τον πυρισμό των εργασιών μεταξύ του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και του Συμβουλίου Εξωτερικών. Ε, τι διευθετήσεις έχετε. Μετά οι συμφωνίε πλαίσια που έχουν υπογραφεί μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Πάολο Ρανζέλη ήταν ο διαπραγματεύτη Για να το πω ήπια, το Συμβούλιο δεν ήταν πολύ ικανοποιημένο. Ε, υπάρχουν εξελίξει σε αυτό το μέτωπο. Αφού έχετε αναλύσει το θέμα διεξοδικά, έχετε διαφορετική στάση ή πιστεύετε ότι θα έπρεπε ε, να καταλήξει υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σας ευχαριστώ. Κύριος Μπρόνς, ευχαριστώ Πρόεδρε. Μιλήσατε για αλλαγές στη συνθήκη που θα εφαρμοστούν ε, γρήγορα και με απλουστευμένη διαδικασία. Όπως ξέρετε αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί η κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι θα οργανώσει δημοψήφισμα σε περίπτωση αλλαγών που οδηγούν σε εκχώρηση κυριαρχίες. Ελπίζω ότι η απλουστευμένη διαδικασία δεν θα αποβεί βάρος σωστή συζήτηση σε όλες τις χώρες για όλες τις μελλοντικέ αλλαγές. Μιλήστε για επέκταση της οικονομικής διακυβέρνησης. Προποθέτει έλεγχο των προϋπολογισμών και των κρατών μελών. Θεωρείτε κύριε Υπουργέ ότι είναι σκόπιμο για χώρες όπως η Ουγγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο που είναι εκτός Ευρωζώνης να υποστούν παρόλα αυτά έλεγχο του εθνικού τους προϋπολογισμού. Σε ό,τι αφορά το δημοκρατικό έλλειμμα, συμμερίζεστε την ελπίδα μου ότι το εμπόδιο για τη, με τη συμμόρφωση των ευρωπαϊκών αξιών δεν θα χρησιμοποιηθεί ως ε, πρόσχημα για ε, αύξηση των διαφωνιών. Επίσης, ε, αναφέρθηκατε σε πιθανό χρονοδιάγραμμα για την προσχώρηση της Κροατίας. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει και ένα λεπτό τεχνικό ζήτημα που αφορά το δημοψήφισμα που σε αντίθεση με την πρωτοβουλία των πολιτών είναι ένα πραγματικό, ένα γνήσιο παράδειγμα άμεσης δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι η Ουγγαρία για πρώτη φορά ασκεί την Προεδρία. Ξέρετε, εγώ γεννήθηκα την περίοδο του αγώνα του Ουγγρικού λαού για την ελευθερία. Και θυμάμαι αυτά τα οποία είχε πει ο Ούγκρος πρόεδρος όταν είχε ανοίξει το σιδηρούν παραπέτασμα και βρέθηκαν τότε συγγενείς μου στο γραφείο μου στη Βόνη και το τι είχε κάνει τότε η Ουγγαρία. Θα ήθελα να σας πω λοιπόν πως το Κοινοβούλιο έχει επενδύσει πάρα πολύ δουλειά ε, στη συνθήκη της Λισαβόνας για να τεθεί μάλιστα ενισχύτως το μόνο δυνατόν και να είναι διαθέσιμη στους πολίτες της Ευρώπης και μάλιστα η εμπειρία μας τότε από τις διαπραγματεύσεις ήταν πως χρειαζόταν επιγόντως κάποιο στο Συμβούλιο ο οποίος ε, θα παρακινήσει τα, τα κράτη-μέλη. Τώρα θα γίνει το ίδιο και στην ε, εφαρμογή. Και βεβαίως οι εμπειρίες ε, που έχουμε μας λένε πως καλό θα ήταν να βοηθήσει λίγο η Ουγγρική Προεδρία για να φροντίσουν να κάνουν τα κρατημέλη αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν. Επίσης εκεί όπου υπάρχει ακόμα περιθώριο θα πρέπει να είμαστε όσο δυνατόν λιγότερο γραφειοκρατικοί και πιο κοντά στον πολίτη. Να αναφέρω ένα δεύτερο σημείο το θέμα του, της ομπρέλας προστασίας, του Συμφώνου Σταθερότητας ε, και της οικονομικής διακυβέρνησης και θα το διατυπώσω ως ερώτηση. Δεν θεωρείτε... Να, να το πω έτσι. Ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι για τους οποίους δεν θα πρέπει να ακολουθήσουμε την κανονική διαδικασία αναθεώρησης της συνθήκη και θεωρείται πως ειδικά με, αυτές τις, με αυτό το πάρα πολύ επίγον αλλά και δύσκολο, περίπλοκο θέμα δεν θα έπρεπε να έχουμε μια διακυβερνητική διάσκεψη και μια συνέλευση με πολλούς συμμετέχοντες για να έχουμε ακριβώς μεγαλύτερη νομιμοποίηση στα κράτη-μέλη και στους λαούς μας για να έχουμε και λίγο έτσι πιο σοβαρές ε, σκέψεις και μακροπρόθεσμες και να μην τρέχουμε συνέχεια να επιβάλλουμε μέτρα ad hoc που πάλι θα αποδειχθεί πως δεν θα λύσουν σε βάθος χρόνου το πρόβλημα. Περιοριστώ σε αυτά. Είχα και τρίτο θέμα, αλλά βλέπω το ρολόι τώρα και... Σας ευχαριστώ κύριε Χεφνέρ. Τελευταία παρέμβαση από τον κύριο Ράγκελ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ την Ουγγρική Προεδρία όχι μόνο για τους λόγους που ακούσαμε ότι είναι μια χώρα που από απολυταρχικό καθεστώς ασπάστηκε ε, τη δημοκρατία αλλά και για ιστορικούς λόγους που είναι πολύ σημαντική γιατί όπως και η, ε, η Πολωνία, η Ουγγαρία είχαν μια πολύ δύσκολη κατάσταση στην ε, ευρωπαϊκή ε, επικράτεια και τώρα θα έχουν την ευκαιρία να προεδρεύσουν, να πρωτοστατήσουν στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, ε, ότι η Ένωση μας, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει αυτή τη δυνατότητα να φέρνει κάθε φορά έναν λαό και ένα κράτος ε, στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας ε, ευχηθώ καλή επιτυχία, επιτυχία αντίστοιχη με αυτή που έχουν ε, η κυρία Γκουρμάη, ο κύριος Σέπφλιν, ο κύριος Σάιερ, οι Ούγγροι δηλαδή ευρωβουλευτές. Γιατί αν η Ουγγρική Προεδρία έχει αντίστοιχε λαμπρέ επιδόσει με του Ούγγρου Ευρωβουλευτέ, πραγματικά η επιτυχία τη θα είναι εντυπωσιακή. Θα ήθελα να υποβάλω δύο, δύο ερωτήσεις. Τη μία την ε, έκανε και ο κύριος Τροσκόφσκι για την συμφωνία πλαίσιο. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της προσχώρησης νέων μελών. Δεν είπατε τίποτα για την Ισλανδία. Γιατί για λόγους που συνδέονται και με οικονομικά και δημοσιονομικά ζητήματα και θέματα οικονομικής διακυβέρνησης, θα ήθελα να μάθω την άποψη της Ουγγρικής Προεδρίας ως προς την ένταξη της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τώρα την προσχώρηση της Κροατίας, θα πρέπει να είμαστε άκρος προσεκτικοί και συνετοί. Μάλιστα, αυτό φάνηκε και στην τελευταία έκθεση που εγκρίναμε στην Ολομέλεια του Στρασβούργου. Πολύ προσεκτικοί θα πρέπει να είμαστε ως προς τη σχέση μας με τη Σερβία και το θέμα του κοσυφοπεδίου. Φυσικά η Κροατία αξίζει μια καταφατική απάντηση, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε το θέμα της ισορροπίας στα Βαλκάνια. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε μια στρατηγική ένταξης, προσέγγισης ε, και προς τη Σερβία, αλλά και μια προσέγγιση ότι αφορά το θέμα του κοσυχοπεδίου. Η Ουγγρική Προεδρία, που είναι ε, ένθερμη υποστηρίκτρια της προσχώρησης της Κροατίας. Πώς αντιμετωπίζει τις σχέσεις με τη Σερβία και για το θέμα του κοσυφοπαιδίου, γιατί είναι ζητήματα αλληλένδετα που θα ε, τεθούν και συνδέονται και με το θέμα της ένταξης της Κροατίας. Ευχαριστώ. Σταματήσαν οι παρεμβάσεις. Δεν ξέρω αν θέλει η κυρία Γκέωρ να μιλήσει. Διαφορετικά, η θα δώσω το λόγο στον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Έχετε το λόγο. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις άκρως ενδιαφέρουσες σχετικές ερωτήσεις και σχόλια που ακούστηκαν. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάθε ένα από αυτά που ετέθησαν, συνδυάζοντας ενδεχομένως μία, δύο, τρεις ερωτήσεις που αφορούσαν το ίδιο θέμα, για να επιταχύνω και να διευκολύνω και το έργο των διαρμηνέων δεν θα αλλάζω γλώσσες. Θα απαντώ στη γλώσσα, στην... Ε, ανεξάρτητα το σε ποια γλώσσα το ερώτημα, θα απαντήσω αγγλικά γιατί ξέρω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Η Κροατία τώρα. Ναι. Έχει τεθεί σαφώς ότι θέλουμε να ολοκληρώσουμε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Κροατία μέχρι το τέλος της Ουγγρικής Προεδρίας. Αυτό δεν σημαίνει υπογραφή τη συμφωνίας. Αυτό μπορεί να ακολουθήσει. Ελπίζουμε κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας. Πριν το τέλος ενεστώτος τρέχοντος έτου. Αλλά κυρίω μετά την 22 Δεκεμβρίου όπου τρία συμπροματικά κεφάλαια έκλεισαν όλοι οι ειδικοί λένε ότι έχουμε αρκετές πιθανότητες ε, ότι μπορούμε να καταφέρουμε αυτό που προανέφερα. Δεν ξέρω αν θα πραγματοποιηθεί η πρόβλεψη ή όχι. Αυτό που λέμε σαφώς είναι ότι είναι μία από τις προτεραιότητές μας, τους στόχους μας. Απομένουν επτά κεφάλαια, δεν είναι ο αριθμός που μετράει, αλλά τα ζητήματα τα οποία καλύπτονται. Όλοι γνωρίζουν ότι το κεφάλαιο 23 είναι κρίσιμη σημασία. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να τοποθετηθεί τον Μάρτιο Εκεί θα είναι αποφασιστικός ο παράγων κατά πόσο θα μπορέσουμε να κλείσουμε το κεφάλαιο 23 και κάτι άλλο βέβαια. Η συνεργασία με το ICTI, εκεί είμαι πιο φιλόδοξος. Το ποινικό δικαστήριο της Χάγης, ελπίζουμε όλα να γίνουν, να πάνε κατευχήν και αυτός είναι ο στόχος μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Γιώζεφ. Σε ευχαριστώ για τα προσωπικά σου σχόλια. Uh, I uh, of course, uh, reflect upon that. Θα το σκεφτούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που μου ήρθε στο μυαλό ότι είναι πράγματι η πρώτη φορά που τίθεται το θέμα. Την επόμενη φορά που αναλαμβάνουμε την Προεδρία, σε 14-15 χρόνια θα επανακάμψουμε στην Προεδρία. Εξαρτάται πόσες νέες χώρες θα ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία που έχουμε, διότι είναι, είναι ιδιαίτερη χάρη αυτή που μας δίνει η ιστορία. Ε, κύριε Νταφ, το συζητήσαμε αυτό συντομία στη Βουδαπέστη και Από ό,τι κατάλαβα, και από την πλευρά της οικονομικής σταθερότητας, αυτή η αναθεώρηση της συνθήκης δεν αρκεί. Πιστεύω, και απαντώ εδώ και σε άλλα που υπόθηκαν, ότι αυτό είναι εκείνο που μπορούμε να κάνουμε τώρα. Στην παρούσα οικονομική, στο παρόν οικονομικό και χρηματοπιστωτικό κλίμα πιστεύω ότι το εγχείρημα θα πρέπει να είναι περιορισμένη εμβέλεια και να είναι γρήγορη προσπάθεια. Δεν έχουμε μόνο 27 παίκτε. δεν έχουμε μόνο το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά έχουμε κι άλλον ένα παίκτη στο παιχνίδι, τις αγορές και δεν αναφέρομαι στην κοινή γνώμη των χωρών. Αν τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη, πιστεύω ότι η προσπάθειά μας θα πρέπει να είναι περιορισμένη και ταχεία. Ιώζεφ, συγγνώμη, ξέχασα το ερώτημά σου. Για τους ε, πίνακες συσχετισμών σε διαβεβαιώ ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ούτω ώστε αυτοί οι πίνακες να ετοιμαστούν σωστά. Το κάναμε οι ίδιοι. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Δεν θέλω να κατηγοριοποιήσω τα κάτι μελη δεν θέλω να, να τα διαχωρίσω τα κάτι μελη μεταξύ παλαιών και νέων. Έχουμε ένα κοινό στόχο. Αυτοί οι πίνακες αντιστοιχίες των σχετισμών να ετοιμαστούν και θα είναι σημαντικός μοχλός για τη συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Για την οικονομική διακυβέρνηση θα είναι δύσκολες οι συζητήσεις, οι διαπραγματεύσεις. αρκετά περίπλοκες ε, θα καλυφθούν σημαντικά ζητήματα τα προβλήματα μπορεί να επιληφθούν ο ρόλος των διαφόρων θεσμικών ε, οργάνων ο αυτόματος χαρακτήρας κάποιων διαδικασιών και άλλα τυχόν ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν. Πιστεύω ότι εάν συσχετίσουμε την οικονομική διακυβέρνηση και τη σχετική νομοθεσία και άλλα ζητήματα, με άλλα ζητήματα, τότε ε, δυσκολεύουμε κάπως την προσπάθειά μας. Για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο έγιναν συζητήσεις μεταξύ Κοινοβουλίου, του Προέδρου του Κοινοβουλίου, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ούγγρου Πρωθυπουργού Ανοιχτή ήταν η συζήτηση, μπήκαμε σε κάποια σημεία σε βάθος, επί της ουσίας, και παίρνουμε πολύ στα σοβαρά αυτή τη συνεργασία και την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην προετοιμασία του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. για εκλογικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις σε βαθύτερο επίπεδο. Ξέρετε ποια είναι η απόψή μου κύριε Νταφ. Και υπό την ιδιότητα του Συμβουλίου μπορώ να πω ότι αυτή η ιδιότητα δεν μου επιτρέπει να μπω σε λεπτομέρειες. Προσωπικά λέω ότι θα χαιρόμουν πολύ να συζητούσα το θέμα μαζί σας αμέσως μετά την ε, Ουγγρική Προεδρία. Για την ώρα δεν βλέπω πιθανότητες να μπει στην ημερήσια διάταξη. Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό πρέπει να κάνουμε, αναθεώρηση της συνθήκης όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας κατά τα λοιπά, γνωρίζοντας ότι είναι εξελικτική αυτή η διαδικασία, έχει κρατήσει πάνω από μισό αιώνα, είναι αέναη, δεν ξέρουμε τι μορφή θα έχει στο μέλλον, τα επόμενα χρόνια και δεκαετίες. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι πρέπει να συνεχίσουμε. Το πώς θα συνεχίσουμε, με ποια ταχύτητα, υπό ποια μορφή, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Τώρα η πρωτοβουλία των πολιτών... Α, συγγνώμη. Πρώτα απ' όλα η κύρωση της συνθέσεως του Κοινοβουλίου, πολύ σημαντικό, 13 από τα 27 κρατημέλη έχουν κυρώσει. Από αυτά, 7 είναι τα νέα των εισαγωγικών. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και μπορώ να υποσχεθώ στον εαυτό μου είναι να ενθαρρύνουμε όλα τα κρατημέλη μελη ώστε να λάβει η χώρα η κύρωση του ταχύτερο δυνατόν. Χρειαζόμαστε 27 κυρώσεις θα προσπαθήσουμε λοιπόν να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Υπάρχει και θέμα αξιοπιστίας εδώ που τίθεται. Πρωτοβουλία των πολιτών. Να επαναλάβω αυτά που προανέφερα. Πιστεύω ότι είναι σημαντικότατο ζήτημα. Αλλά πατώντα άλλο σχετικό ερώτημα πρέπει να πω ότι δεν νομίζω ότι επιλύεται ο τρόπος το δημοκρατικό έλλειμμα, αυτό που επεκαλεί το δημοκρατικό έλλειμμα. Εδώ μιλάμε για ένα μόνο στοιχείο. Πρέπει να βρούμε τρόπους μέσα με τα οποία η Ευρώπη να γίνει πλέον δημοκρατική. Αυτή είναι μια δυνατότητα. Σε ποιο βαθμό θα χρησιμοποιηθεί είναι ανοιχτό θέμα. Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι πολλοί ήδη με προσέγγισαν εμένα τον ίδιο. Τι τελευταίε εβδομάδε και μήνε μου είπαν μπορούμε να το κάνουμε τώρα, να ξεκινήσω τη συλλογή υπογραφών. Ε, Πώ πάει το πράγμα. Μπορεί αυτό το θέμα να, να μπει να τεθεί και εγώ να εξηγήσω, κοιτάξτε αυτό δεν είναι ακριβώς κάτι το οποίο μπορεί να καλυφθεί αυτή τη δυνατότητα. Άρα ο κόσμος το γνωρίζει και περιμένει ο κόσμος. Και συμφωνώ με όλου όσοι είπαν ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να επιταχυνθεί και αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να δοθεί μετά την επίλυση όλων των τεχνικών δυσκολιών να ενθαρρυνθούν και τα κρατημέλη να κάνουν τη δουλειά τους αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνει τη δουλειά ε, της, για την σύστημα συλλογής υπογραφών κλπ. Οι τεχνικέ δεπτομέρειε πρέπει να επιληθούν και ταχύτερο δυνατόν θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Ή σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, πώς προβλέπει ο κανονισμός ο σχετικός. Το Σύνταγμα. Να πω ένα-δύο πράγματα, διότι είναι μεγάλο θέμα αυτό. Το Σύνταγμά μας άλλαξε ουσιαστικά Κάποιοι είπαν 95-96-97% όταν άλλαξε το σύστημα. Ο τίτλος του συντάγματος είναι πράξη παριθμών 20 του 1949. 1949 ξέρετε ότι ήταν η χειρότερη χρονιά εκτός από το 44 για τη χώρα μου. Άρα είναι παράλογο να έχουμε τέτοιο τίτλο. Εν πάση περιπτώσει, πολλές προσπάθειες έχουν γίνει για την υιοθέτηση νέου συντάγματος. Ξεκίνησαν οι προσπάθειες το 1994. Εγώ ίδιος είχα συμμετάσχει στην ε, προσπάθεια. Ήταν σοσιαλιστική φιλελεύθερη κυβέρνηση. Κάναμε πρόοδο κατά τη διάρκεια της τετραετίας, σημαντική πρόοδο, άλλαξε η κατάσταση και πάλι και τώρα συνεχίζουμε την ε, όλη προσπάθεια, αυτή τη δουλειά και νομίζω κύριε Γκερέρο ότι η έκφραση που χρησιμοποίησατε ότι έπρεπε εγώ να χρησιμοποιήσω και τις δύο ιδιότητες και τα δύο καπέλα ταυτόχρονα είναι η καλύτερη πρόταση και θέλουμε να την ακολουθήσουμε. Την ακολουθούμε. Τι κάνουμε δηλαδή. Τη χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων αυτολεξεί την εντάσσουμε στο νέο Ουγγρικό Σύνταγμα. Ενώ είναι κοινοτική νομοθεσία για τον τομέα στον οποίο εφαρμόζεται, παρόλα αυτά θα αποτελεί τμήμα του Ουγγρικού δικαίου και θα είναι εφαρμοστέο σε κάθε τομέα. Αυτό είναι το μέγιστο που μπορούμε να κάνουμε. Άρα, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα τα συμπεριλάβουμε στο Σύνταγμα και το Σύνταγμα θα έχει ενσωματωμένη την Ευρωπαϊκή Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ήδη αναφέρθηκα ακροθυγός στη διεύρυνση, στο ζήτημα της διεύρυνσης που ετέθη από την κυρία Λεγκρή. Γνωρίζετε τι γίνεται με το σκεπτικισμό, υπάρχει διστακτικότητα και πρέπει να σεβαστούμε και την αρχή της αιρεσιμότητας. Ας μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Από τη μία πλευρά προσπαθούμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και να τις ενθαρρύνουμε, ταυτόχρονα όμως πάντα λέμε στις υποψήφιες χώρες ότι και αυτές θα πρέπει να κάνουν αυτό που τους αρμόζει. Δύσκολα να, να ετοιμάσουμε χρονοδιάγραμμα, σε κάποιους δεν αρέσει καθόλου, διότι πιστεύουν ότι οι ημερομηνίε πρέπει να επιλέγονται προσεκτικότατα, όμως νομίζω ότι η ώρα της αλήθειας θα φτάσει. Όταν ξεκινήσουμε δηλαδή τη συζήτηση βασικών θεμάτων του προπολογισμού θέματα χρηματοδότησης και συνοχής και της σχετικής πολιτικής, τότε θα πρέπει να καθορίσουμε ένα θεωρητικό τουλάχιστον χρονοδιάγραμμα για την ένταξη της Κροατίας, η ημερομηνία για την ένταξη της Κροατίας. Δεν πρέπει να λησμονούμε τις άλλες χώρες. Αντιθέτως, αυτό που κάνουμε, αυτό που λέμε είναι ότι αν τα καταφέρουμε με την Κροατία, αν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τι διαπραγματεύσεις με την Κροατία, αυτό θα είναι το καλύτερο μήνυμα που στέλνουμε προ του άλλου. Ότι και εκείνε οι χώρε έχουν επίση τη δυνατότητα, κάποτε θα έχουν δυνατότητα. Η Ουγγαρία κάποτε ήταν από τι πρώτε χώρε, μάλλον που επικύρωσε τη Συμφωνία σταθερότητα με την Σερβία. Ήταν από τι πρώτε χώρε η Ουγγαρία που έλεγε ότι θα έπρεπε να αρχίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προετοιμάσει την ε, γνωμοδότησή της και χαιρόμαστε διότι σε δύο μέρες περίπου η σερβική κυβέρνηση θα υποβάλει συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο όπως αποκαλείται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε θα είναι σε θέση να ετοιμάζει την περίφημη γνωμοδότησή της ή αβή όπως αποκαλείται που είναι πάρα πολύ σημαντική όσον αφορά την ένταξη της ε, Σερβίας. Αξιολόγηση της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Συμφωνώ πλήρως ως προς την ενθάρρυνση αυτής της διαδικασίας και την επιτάχυνσή της. Το είπα και προηγουμένως. Θα πρέπει να προωθήσουμε την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επανέρχομαι τώρα στα σχόλια του George Shepflin. Η πρωτοβουλία των πολιτών είναι ένα μόνο μέσο, ένα μόνο εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας. Αλλά θα χρειαστεί για πολύ καιρό να ασχοληθούμε με τον Ευρωπαϊκό Δήμο και πώς θα προωθήσουμε αυτή την ιδέα του Ευρωπαϊκού Δήμου. Θα σας δώσω ένα απλούστατο παράδειγμα. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες ευρωσκεπτικιστικές τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη και στη δική μου πατρίδα, ε, στην Ουγγαρία, χάρη στην Προεδρία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει πιο δημοφιλής. Δεν ξέρω αν είναι παράδοξο αυτό ή όχι, αλλά υπάρχει εξαιτία τη εξοικείωση ε, που αποκτά ο Ουγγρικό λαό ε, μέσω τη Προεδρία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, φαίνεται να αυξάνεται η υποστήριξή του προ αυτή. Υπάρχει περισσότερη αφύπνιση και καλύτερη συνειδητοποίηση και προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ την Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη. Το θέμα των ε, αλλαγών στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Ήταν ένα ζήτημα που απασχόλησε πολλούς ευρωβουλευτές στις παρεμβάσει του Θα ήθελα απλώ να επαναλάβω ότι η Ευρωζώνη είναι μια πραγματικότητα, αμετάβλητη. Αν θέλουμε λοιπόν να θεσπίσουμε για τις ζώνες της Ευρωζώνης έναν μηχανισμό σταθερότητας, ένα είδος μηχανισμού διάσωσης που θα στηρίζεται σε συνεισφορές των χωρών της Ευρωζώνης, αυτό θα γίνει μόνο από τα μέλη της Ευρωζώνης. Μόνο αυτά μπορούν να αποφασίσουν και να θεσπίσουν ένα τέτοιο μηχανισμό. Φυσικά εμείς μπορεί ad hoc, αν παραστεί ανάγκη, να προσχωρήσουμε, αλλά δεν μπορούμε εμείς να παρέμβουμε στους κανονισμούς και τους κανόνες για τις αρμοδιότητες των μελών της Ευρωζώνης όπως αναφέρονται στις συνθήκες. Το θέμα της κύρωσης βέβαια είναι επίσης σημαντικό. Αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που συντρέχουν υποθέσεις για την απλουστευμένη διαδικασία δεν υπάρχει καμία εκχώρηση αρμοδιοτήτων. Είναι θέμα 3. Πιστεύω ότι μπορούμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία αυτή για την έγκριση αυτών των αλλαγών. Νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα που θα στείλουμε και προς την κοινή γνώμη. Αλλά και ένα χειρό μήνυμα προς τις αγορές. Σε ό,τι αφορά την οικονομική διακυβέρνηση, όπως είπα, το θέμα αυτό είναι ξεχωριστό και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Δεν νομίζω ότι ένα είδος ελέγχου των προϋπολογισμών παραβιάζει ή παρεμβαίνει στην κυριαρχία των κρατών μελών. Αυτό τα λέει, το προβλέπει η συνθήκη. Και η νομική βάση για τα έξι νομοθετικά κείμενα ήδη υπάρχει στη συνθήκη. Γιατί μιλούμε για συντονισμό των οικονομικών πολιτικών αυτά τα θέματα ήδη κατοχυρώνονται ήδη και Παρόλο που ακόμη ο συντονισμό αυτό δεν έχει γίνει πραγματικότητα στην έκταση που θα περιμέναμε. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να επικεντρωθούμε στο θέμα της οριστικοποίησης και της ολοκλήρωσης αυτών των έξι νομοθετικών κειμένων. Ένα τελευταίο θέμα, πολύ σημαντικό όμως, είναι ότι φυσικά είμαστε υπέρ της ένταξης της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλλον θα έχουμε τον πρώτο γύρο των πρωταξιακών διαπραγματεύσεων κατά το τέλος της Ουγγρικής Προεδρίας αλλά αυτή φυσικά θα είναι αφετηρία και όχι διεκπαιρέωση της διαδικασίας θα τη συνεχίσουν ε, οι Πολωνοί συνάδελφοι η επόμενη Προεδρία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πολωνό συνάδελφο για τις παρατηρήσεις τους. Πραγματικά είναι μια ιστορική σημασία, σε ευκαιρία για μας και τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Θα είναι πραγματικά το 2011 το έτος της Κεντρικής Ευρώπης. Θα έχουμε τρία διαφορετικά τρία, αλλά σίγουρα θα έχουμε και σε αυτό και στο επόμενο τρίο χώρες Κεντρικής Ευρώπης. Και ευελπιστώ ότι θα είναι και τυχερό και επιτυχημένο αυτό το ημερολογιακό έτος για όλους μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για άλλο το χρόνο που μας διαθέσατε σήμερα το πρωί και για τις ακριβείς απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις μας. Μπορούμε σε αυτό το στάδιο να σταματήσουμε τη συνάντηση μαζί σας, αναδιατυπώνοντας ξανά τις ευχές μακάρι να είναι ακρογωνίως λήθος η ε, Ουγγρική Προεδρία στη διαδρομή της Ευρώπης προς μια μεγαλύτερη ολοκλήρωση. Ελπίζουμε και ευχόμαστε η Ουγγρική Προεδρία να ε, εγγραφεί στην ιστορία σαν ποιοτικό άλμα στην ε, διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και θα πάμε τώρα στην ακρόαση όσον αφορά τα πολιτικά κόμματα. Ας διακόψουμε για δύο λεπτά τη συνεδρίαση, ώστε να χαιρετήσω και τον κύριο Υπουργό. Ξεκινάμε λοιπόν το δεύτερο τμήμα. Ξεκινάμε το δεύτερο τμήμα της συνεδιάσεώς μας που αφορά την εφαρμογή του κανονισμού 2004-2003 για το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή η μερίδα είναι αφιερωμένη σε αυτό το θέμα και θα κατανεμηθεί σε τρία τμήματα. Σήμερα το πρωί θα ακούσουμε προσωπικότητες που ηγούν των διαφόρων ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Όπως γνωρίζετε, το άρθρο 10 της Συνθήκης της Ένωσης δηλώνει ότι τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμβάλλουν στο δημιουργηθεί μια συνείδηση πολιτική ευρωπαϊκή και να εκφράζουν τη βούληση των ε, πολιτών της Ένωσης. Ο κανονισμός μας που παρέθεσε 2004 του 2003 ρυθμίζει το καθεστώ και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προβλέπεται στον κανονισμό μεταξύ άλλων ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάσει μια έκθεση που αφορά την εφαρμογή αυτού. Θελήσαμε λοιπόν να διοργανώσουμε κατόπιν ετήματος τη εισηγήτριάς μα, τη κυρία Γιαννάκου, αυτή την ακρόαση για να συζητήσουμε ε, τα προβλήματα να ακουστούν προτάσεις και να γίνουν αξιολογήσεις και εκτιμήσεις πέραν από το προσωπικό των πολιτικών κομμάτων που είναι παρόντα εδώ τα μέλη αυτά. Έχουμε την ακρόση των πυρογνωμών το απόγευμα, καθηγητών πάνω στο θέμα αυτό και πιο συγκεκριμένα σήμερα το βράδυ θα παρουσιαστεί μια μελέτη όσον αφορά τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα ε, υπερεθνικό ε, πολιτικό σύστημα και θα ακούσουμε το απόγευμα τον εκπρόσωπο του ελεκτικού συνεδρίου όσον αφορά τις οικονομικές πτυχές για τα κόμματα και εκπρόσωπο ε, που θα αναφερθεί στην ε, διεθνή διαφάνεια. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις θα μας επιτρέψουν, θα επιτρέψουν στους βουλευτές, τα μέλη της Επιτροπής μας, να εκφράσουν την άποψή τους, να υποβάλουν ερωτήσεις και στην κυρία Γιαννάκου να κλείσει τη σημερινή συνεδρίαση. Το πρωί ακούσαμε τους, θα ακούσουμε τους εκπροσώπους μάλλον των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων. Δυστυχώς, λόγω περιορισμένου χρόνου, δεν μπορώ να επιτρέψω παρά μόνο πέντε λεπτά σε κάθε προσωπικότητα. Ίσως εκείνοι που πρέπει να παρέμβουν Εάν μιλήσουν, θέλουν να μιλήσουν πολύ, ίσως να μειώσουμε ακόμα περισσότερο το χρόνο στα μισά ε, για να ακούσουμε τις παρεμβάσεις των μελών της Επιτροπής. Και στα μισά της ε, να ακουστούν οι απόψεις τους στις συνομιλίες. Η πρώτη προσωπικότητα λοιπόν που θα πάρει το λόγο είναι πρόεδρος Μάρτενς και δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις στο Κοινοβούλιο, όμως να επενθυμίσω τα βασικά είναι πρώτη στην πολιτική προσωπικότητα, ήταν πρωθυπουργό μεταξύ 79 και 82 στη χώρα του και ήταν επικεφαλής ε, σοσιαλχριστιανικής φιλελεύθερης ε, ε, συνασπισμού μάλλον. Δεν πρέπει να επιθυμήσω που ο από τις 10 Μαΐου του 1990 ήταν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ήταν από τους ιδρυτές του κόμματος. Ο Βαλδουίνος ο πρώτος το 1992 του έδωσε το, ε, τίτλο του Υπουργού ε, επίτιμο ε, Υπουργό. Λοιπόν, θα μπορούσα να πω πολλά, αλλά επειδή πρέπει να μιλήσουν οι προσωπικότητε, δεν θα χρονοτριβήσω προ τι συστάσει. Αγαπητέ κύριε Μάρτιν, σα δίνω το λόγο. Thank you very much, Mr. President. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την Επιτροπή σας και το Κοινοβούλιο σας. Έδειξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε ένα από τα κύρια ευρωπαϊκά κόμματα. Ε, έχω πέντε λεπτά. Θα θυμάστε ότι ως ε, Πρωθυπουργό της χώρα μου στι διαπραγματεύσει για τη συνθήκη του Μάστριχτ ανέλαβα την πρωτοβουλία αναγνώρισης και χρηματοδότησης των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων. Ήμασταν τότε 12 πρωθυπουργοί, ήταν το πρώτο θέμα της μερίσιας διάταξη. και μετά από συζήτηση 50 λεπτών έγινε δεκτό το Δεκέμβριο του 1991 και μετά στη συνθήκη του Μαστρίχτ είχαμε το διάσημο άρθρο 138α τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σημαντικά ως παράγοντες ενοποίησης εντός της Ένωσης. Και θα θυμάστε κύριε Πρόεδρε τη φράση συνεισφέρουν στην διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής συνείδησης και στην έκφραση της πολιτικής βούλησης των πολιτών της Ένωσης. Έχω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, η πρώτη φράση, τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σημαντικά ως παράγον ενοποίησης εντός της Ένωσης, εξαφανίστηκε στο άρθρο 14 της Συνθήκης της Λισαβόνας και η δεύτερη παρατήρηση είναι πως δεν υπήρχε αναφορά για τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Χρειάστηκαν 13 χρόνια από το 1992 την συνθήκη του Μαστρίχτ. Όχι. 8 χρόνια μέχρι την ε, συνθήκη της Νίκαιας και το άρθρο 191 για να γίνει αναφορά σε χρηματοδότηση. Γιατί ήταν ουσιώδες αυτό για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Χρόνια και χρόνια ζούσαμε από τις συνεισφορές των ε, κομμάτων μελών. Αλλά ήταν σημαντικό να είμαστε πιο αυτόνομοι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανεξάρτητοι και να έχουμε τα απαραίτητα μέσα για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Χρειάστηκαν μάλιστα 13 χρόνια πριν να δοθεί αυτή η χρηματοδότηση. Και στο ψήφισμα αυτό, την απόφαση αυτή και με τη χρηματοδότηση αυτή και την αναγνώριση όπως είπα έπαιξε σημαντικό ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην έκθεση Λάγκεν είχαμε μια αναθεώρηση και θα επανέλθω σε αυτή. Και στην έκθεση του κυρίου Λάινεν είπε πως δεν χρειαζόμαστε μόνο τη χρηματοδότηση και ήταν λύση για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα αλλά είπε επίσης στην έκθεσή του τόνισε την ανάγκη για ένα πραγματικό ευρωπαϊκό καταστατικό κομμάτων που πηγαίνει πέρα από τη χρηματοδότηση κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ζήτησε να έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις και το δικαίωμα να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα βασισμένη στο κοινοτικό δίκαιο με υπόσταση στα κράτη-μέλη και ζήτησε να σκεφτεί η Επιτροπή σας το ζήτημα ευρωπαϊκού καταστατικού από και οικονομική σκοπιά και να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για το σκοπό αυτό. Οπότε, παραλαμβάνω, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για τη χρηματοδότηση, αλλά αυτή δεν είναι πλήρης αναγνώριση. Χρειαζόμαστε νομική και πολιτική νομιμοποίηση για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και υπάρχουν πολλές σημαντικές προτάσεις για να τονίσουμε αυτή την νομοποίηση και αυτό είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε παραδείγματος χάρη για την ευρωπαϊκή πολιτική συζήτηση παραδείγματος χάρη για τον ορισμό υποψηφίων ε, για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παραδείγματο χάρη, και αναφέρομαι εδώ πέρα στην έκθεση DAF, για να δημιουργηθεί λίστα πανευρωπαϊκή. Τώρα είμαστε μη κερδοσκοπικές ενώσεις. Στις ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες ε, ε, υπάρχουμε. Δεν έχουμε λοιπόν το νομικό και πολιτικό καθεστώς που θα μας επιτρέψει να παίξουμε πραγματικό πολιτικό ρόλο. Και ελπίζω και ευχαριστώ ειδικά και τον εισηγητή, την εισηγήτρια για τις ερωτήσεις της. Ελπίζω το επόμενο βήμα σε αυτή την συζήτηση και μετά την ε, δημόσια κρόση και αφού ακούσουμε τους ειδικού να είναι να κάνουμε το παραπέρα βήμα για να δημιουργήσουμε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Λάινε στην έκθεσή του αυτό το πολιτικό και οικονομικό και φορολογικό καθεστώς για τα πολιτικά κόμματα. Το μέλλον επίσης και φορολογικό καθεστώς να βρούμε μία λύση η generis. Καταλήγοντας, για τα ερωτήματα και τις προτάσεις του Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμφωνούμε, νομίζω πως έχει ξεχάσει τα συμπεράσματά του, πως για την αναγνώριση κάθε Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα θα πρέπει να εκπροσωπείται από τουλάχιστον έναν Ευρωβουλευτή είναι αυτό στα, σε σκέψεις και όχι στα συμπεράσματα του Γενικού Γραμματέα, αλλά για μένα είναι ουσιώδες. Στις προτάσεις αυτές αποδέχεται τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και από τα περιφερειακά κοινοβούλια, αλλά ουσιαστικό είναι να έχουμε ερετούς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και λέει σε αιτιολογικές σκέψεις πως τουλάχιστον ένας ευρωβουλευτής είναι κάτι το αναγκαίο για να υπάρχει αναγνώριση Ευρωπαϊκού Πολιτικού Κόμματος. Οπότε αν θέλουμε πράγματι πολιτικά κόμματα στο πνεύμα της ομοφωνίας των διαπραγματεύσεων του Μάστριχτ που ανέφερε πώς θα παίξουν αυτό το ρόλο το σημαντικό για την ολοκλήρωση της Ένωσης, χρειαζόμαστε αυτό το βήμα και ελπίζω τώρα να είστε ανοιχτοί, διατεθειμένοι για αυτές τις συζητήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν την κατάληξη ναι. αυτού του έργου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και όλα τα μέλη της Επιτροπής σας. Σας ευχαριστώ κύριε Μάρτινς. Δίνω το λόγο στο Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Συστικού Κόμματος τον κύριο Φιλίπ Κορντερή, ο οποίος το 2004 είχε αναλάβει τα καθήκοντά του και είχε πολλά καθήκοντα εντός του Σοσιαλιστικού Κόμματος, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου από το 1994 του Σοσιαλιστικού Κόμματος και ήταν και διεθνής γραμματέας του Κινήματος των Νέων Σοσιαλιστών, των Γάλλων, από το 1990 και ήταν και στο γραφείο του Προέδρου της Γαλλικής Συνέλευσης μερικές πινελιές εδώ για να σας δείξω πόσο σημαντικό πρόσωπο είναι και σας δίνω το λόγο τώρα. Έχετε το λόγο κύριε Φιλίπ Κορντερή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρου του Πολ Νίροπ Ράσμουσεν, του Προέδρου του ε, Σοσιαλιστικού Κόμματο. Κανονικά εκείνο έπρεπε να είναι, αλλά δημιουργήθηκε μια σύγχυση και έτσι τον αναπληρώνω εγώ σήμερα. Σα ζητώ συγγνώμη εκ μέρου του. Επίση, θα ήθελα επί ευκαιρία να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, την εισηγήτρια, αλλά και τα μέλη του Προεδρείου, ε, τον κύριο Λαμπρινίδη, που στο Προεδρείο, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα, κατέθεσαν την πρόταση που εξετάζουμε σήμερα και μπορούμε να την αναπτύξουμε. Ο πρόεδρος Μάρτενς ε, μας περιέγραψε πολύ σωστά την πρόοδο που σημειώσαμε στο θέμα του Ευρωπαϊκού Πολιτικού Κόμματος ε, και οι εξελίξει από το 2004 και μετά μας επιτρέπουν να έχουμε σήμερα κάποια κόμματα που αρχίζουν να έχουν μία ζωή αλλά και μία επιρροή στην ε, ευρωπαϊκή πολιτική συζήτηση. Σήμερα όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να πολιτικοποιήσουμε πολύ περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιτρέψουμε στον πολίτη να αντιληφθεί καλύτερα τις ευρωπαϊκές προκλήσεις και τα διακυβευόμενα και να παρακολουθήσει τις διάφορες ε, προτάσεις που εξετάζονται στην Ευρώπη. Θα πρέπει οι Ευρωπαίοι πολίτε να αντιληφθούν ότι οι ευρωπαϊκέ προκλήσει είναι εξίσου σημαντικέ με τις τοπικές και τις εθνικές και να αντιληφθούν του διαφορετικούς πολιτικούς προσανατολισμούς και το πώς τους εκπροσωπούν τα διάφορα κόμματα. Η δημοκρατία είναι ένα κοινό θεμέλιο για όλους μας και όλοι όσοι συμμετέχουμε εδώ στην Ομίγυρη γνωρίζουν ότι σε όλες τις εθνικές δημοκρατίες τα πολιτικά κόμματα διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο και αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του δημοκρατικού βίου μιας χώρας. Οπότε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σημαντικό να, να πραγματοποιήσουμε αυτό το ποιοτικό άλμα πρόοδου και να έχουμε πραγματικά ε, ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα που θα διαδραματίζουν σωστά το ρόλο τους, που θα είναι αντίστοιχο με των ε, εθνικών πολιτικών κομμάτων στα πλαίσιο των εθνικών δημοκρατιών. Στις τελευταίες ευρωεκλογέ ε, είδαμε τι ρόλο μπορούν να έχουν τα κόμματα με το ισχύον καταστατικό. Όλοι ε, εκδώσαμε σημαντικά μανιφέστα, είχαμε πολύ σημαντικές δράσεις της ε, εκστρατείας, αλλά παρόλα αυτά οι, εκστρατείες, οι προεκλογικές εκστρατείες δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν τον εθνικό κλειό, την εθνική διάσταση, ώστε να έχουμε πραγματικά ευρωπαϊκές συζητήσεις με, ε, μεταξύ πραγματικών γνήσιων ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Και αυτό χρειαζόμαστε με το νέο καταστατικό. Μιλήσαμε για μια νομική οντότητα, Μιλήσαμε για σημαντική πρόοδο που πραγματοποιήθηκε σε φορολογικό αλλά και σε επίπεδο χρηματοδότηση, αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να μείνουμε στο πολιτικό ρόλο αυτών των κομμάτων. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να έχουμε εκστρατείε ω ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, να μπορούμε να έχουμε αναγνωρισμένους υποψηφίους στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, από το 2014 για τις εκστρατείες, να έχουμε διακρατικούς ε, καταλόγους υποψηφίων, να μπορούμε και εμείς ε, να πραγματοποιούμε ενημερωτικές εκστρατείες όταν γίνονται δημοψηφίσματα και να μπορούμε να προσφέρουμε και την πολιτική υποστήριξη, όχι χρηματοδότηση, γιατί ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνει και το Συμβούλιο, οπότε είναι σημαντικό να συμμετέχουμε στις στους διάφορους πολιτικούς σχετισμούς που διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως είπε και ο πρόεδρος Μάρτινς, είναι σημαντική η συμβολή των πολιτικών κομμάτων και καλό θα είναι να συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις και να έχουν τακτικές επαφές με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επηρεάζουν τους προσανατολισμούς της ευρωπαϊκής πολιτικής. Νομίζω ότι μπορούμε πολλά περισσότερα να προσφέρουμε ως αναγνωρισμένα πολιτικά κόμματα με συγκεκριμένο καταστατικό. Θα πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός που σήμερα αφορά τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Χρειαζόμαστε ένα κανονισμό για την οργάνωση και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Όχι ένα κανονισμό που απλώς θα προσδιορίζει τις επιδοτήσεις, αλλά θα προβλέπει ταυτόχρονα και μια πολιτική οργάνωση των κομμάτων αυτών. Σήμερα το νομικό μας ε, καθεστώς ε, είναι αντίστοιχο με μιας βελγικής ε, μη Κυβερνητική οργάνωσης. Δεν μας ικανοποιεί αυτή η κατάσταση. Χρειαζόμαστε ένα ειδικό καθεστώς για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και συμφωνώ απόλυτα με τον προλαλήσαντα, τον πρόεδρο του ΕΛΚ, ότι χρειαζόμαστε τουλάχιστον έναν ευρωβουλευτή. Αυτό είναι το, η ελάχιστη προϋπόθεση, απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Πολιτικού Κόμματος. Αλλά χρειαζόμαστε εκπροσώπους και σε διάφορες χώρες, ώστε πραγματικά αυτά τα κόμματα να, να είναι αντιπροσωπευτικά του, της σκέψης, του ρεύματος σκέψης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν πρόκειται να επισέλθω σε λεπτομέρειες γιατί εξαντλήθηκε ο χρόνος μου. Πάντως, συμμεριζόμαστε τις ιδέες της έκθεσής σας. Έχουμε υποβάλει και γραπτό κάποια σχόλια. Το ουσιώδες πάντως για μας είναι να περάσουμε σε μια επόμενη φάση και να έχουμε ένα πραγματικό πολιτικό και νομικό καθεστώς για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Βλέπω ότι προχωράμε γρήγορα. Χάρη σε εσά τηρούμε το χρονοδιάγραμμα. Παρακαλώ. Τώρα η κυρία συνάδελφος Άνεμι Νίτς να πάρει το λόγο που είναι πρόεδρος των Φιλελευθέρων. Υπενθυμίζω ότι ήταν υφυπουργός και μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Φλαμανδικό Βελγικό Κόμμα των Δημοκρατών και Φιλελευθέρων. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας για τη διοργάνωση της ακροάσεως που μας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιαστούμε περαιτέρω και να εκφράσουμε και την άποψή μας όσον αφορά τα βασικά στοιχεία που εμπεριέχονται στο σχέδιο εκθέσεως της συναδέλφους μας, της ε, κυρίας Μαριέτας Γιαννάκου, την οποία να ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά, την καλή δουλειά που κάνει. Λοιπόν, καταρχάς, να υπενθυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Φιλελεύθερο Κόμμα, το οποίο έχω την τιμή να ηγούμε, ιδρύθηκε το 1976 τρία χρόνια πριν από τις πρώτες άμεσες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έλαβαν χώρα το 1979 και ήμουν ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Φιλελεύθερου Κόμματος έκτοτε. Οπότε είδα την εξέλιξή του, είδα πώς ε, αναπτύχθηκε και πώς σήμερα είναι ένα πλήρες πολιτικό κόμμα το οποίο από το 1976 διοργάνωνε ετησίως συνέδρια και τα συνέδριά μας δεν είναι απλώς ε, συζητήσεις ασύλλογοι για συζητήσεις, αλλά είναι πραγματικά, γίνονται πραγματικός πολιτικός διάλογος, υποβάλλονται σχέδια ψηφισμάτων, ψηφίζονται, τροποποιούνται κλπ. Και έτσι εργαστήκαμε για πάνω από 30 χρόνια. Αυτή είναι μία απάντηση στον, στην εσωτερική δημοκρατική λειτουργία που απαιτείται από ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα. Θα ήθελα τώρα να μπω στις απαντήσεις στις τεθήσεις ερωτήσεις που ετέθησαν από τη συνάδελφό μας την κυρία Γιαννάκου. Είμαστε υπέρ ενιαίου καθεστώτος για ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, διότι επί του παρόντος βασικά αντιμετωπίζουμε καμιά φορά αντιφάσεις όσον αφορά τις προϋποθέσεις που υπάρχουν για το νομικό μας καθεστώς σύμφωνα με το βελγικό νόμο. Είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση και κάποιες απαιτήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την οικονομική διοργάνωση και συζητήσαμε το θέμα και με τις βελγικές φορολογικές αρχές που αμφισβήτησαν των τρόπων με τον οποίο παρουσιάζαμε εμείς τα οικονομικά μας στοιχεία. Οπότε υπάρχει ε, ένας βαθμός ενότητας όσον αφορά το καθεστώς θα ήταν κάτι χρησιμότατο. Δεν είμαι τόσο σίγουροι όσο συνάδελφοί μου ότι το καθεστώς αυτό καθεαυτό, το καταστατικό αυτό καθεαυτό θα έδινε παραπάνω νομιμότητα σε ένα κόμμα. Θα μπορούσε να ισχύσει βέβαια κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι η νομιμότητα είναι κάτι που δημιουργείται εκ των έσω και όχι κάτι που σου ε, δίδεται εκ των έξω. Είτε το αξίζεις είτε όχι. Οπότε δυσκολεύει αυτό την όλη κατάσταση. Γίνεται πιο δύσκολη κατάσταση από ό,τι φαίνεται μια πρώτη ματιά. Να κλείσω, το κόμμα μου είναι υπέρ ε, ενός ενιαίου ε, καταστατικού για τα ευρωπαϊκά ε, πολιτικά κόμματα και πιστεύουμε ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα μέλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύουμε επίσης ότι οι εκπρόσωποι των περιφερειακών κομμάτων από περιφέρειες που έχουν νομοθετική εξουσία θα πρέπει να ε, δίνονται, να ε, γίνονται μέλη ε, των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Όσον αφορά την οικονομική πλευρά, πιστεύουμε ότι θα ήταν καλή πρόταση αν στους ιδίου αν οι ίδιοι πόροι θα πρέπει να βγουν εκτός της απαιτήσεω ότι πρέπει να είναι το 15%, να πάνε από 15% στο 10%, θα ήταν χρήσιμο, θα πρέπει να υπάρχει απέτηση, να υπάρχει ένας, ένα επίπεδο ιδίων πόρων, διότι αυτό υποχρεώνει το κόμμα να έχει στενές σχέσεις με τα κόμματα μέλη, διότι οι σφορές τους αποτελούν ε, το βασικό ποσοστό των ιδίων πόρων ε, των κομμάτων μας. Το κόμμα μου επεξεργάστηκε ένα σύστημα για το να προσχωρούν άτομα ως μέλη και θα ξεκινήσουμε εκστρατεία ε, στατολόγηση των εισαγωγικών, προσλήψεως των εισαγωγικών και να δούμε κατά πόσο θα είναι επιτυχές, διότι πιστεύω ότι όλοι οι ορμοί για να γίνουν μέλη, να γίνουν ιδιώτες μέλη ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων δεν είναι τόσο μεγάλη όσο ήταν εδώ και κάποια χρόνια. Αυτός δεν είναι λόγος όμως να το απορρίψουμε ως δυνατότητα, να το προσπαθήσουμε και με τα χαράς να σας τηρούμε ενήμερους σχετικά με την πορεία αυτής της προσπάθειας. Πιστεύω ότι αν θέλουμε όπως υπόθηκε από τους δύο προλαλήσατες, τον πρόεδρο του ΕΡΚ και τον Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, Εάν θέλουμε τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές πολιτικές εκστρατείες, τότε θα πρέπει να επιτρέπεται να ξοδεύουν χρήματα για ευρωπαϊκές πολιτικές εκστρατείες και αυτές οι ευρωπαϊκές πολιτικές εκστρατείες θα είναι πολύ πιο δαπανηρές από ό,τι σε εθνικό επίπεδο, από εθνικές εκστρατείες. Και δεν ε, πρέπει να εθελοτυφλούμε μεταφράζοντας ένα ρητό φλαμαδικό αυτός που λέει α και πρέπει να λέει και β και γ και δ και λοιπά. Αν αυτό το κοινοβούλιο λοιπόν θέλει να δώσει τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές πολιτικές εκστρατείες, τότε θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να μπορούν να διαθέτουν σημαντικά χρηματικά ποσοστά για αυτές τις εκστρατείες. Χρηματικά ποσά μάλλον, συγγνώμη. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο. Απάντησα για τα κομματικά συνέδρια αυτό που είπα για τις πολιτικές εκστρατείες ισχύει επίσης και για τη συμμετοχή μας σε εκστρατείες για δημοψηφίσματα και αν αυτό το κοινοβούλιο αποφασίσει ότι πρέπει να υπάρχει και περιθώριο για υπερεθνικούς καταλόγους θα παίξουμε και εμείς το ρόλο μας για να, να βοηθήσουμε τη δημιουργία των καταλόγων σε ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και αυτό το τελευταίο μου σχόλιο Ήδη έχουμε συμμετάσχει ενεργά και στους διορισμούς των βασικών θέσεων, να το πω έτσι, μετά τις ευρωεκλογέ. Τώρα αν πρέπει να επισημοποιηθεί περισσότερο αυτό στο μέλλον, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε, αλλά θέλουμε σαφώς να παίξουμε το ρόλο μας και σε αυτό το επίπεδο. Σας ευχαριστώ για την ε, προσοχή σας. Ευχαριστώ εσάς, δε Πρόεδρος, κυρία Νέιτς, για... ξέχασα να σας πω ότι ήσασταν μέλος της Επιτροπής μας. Όπως άλλωστε και ο Πρόεδρος ο κ. Μάρτινς και η κυρία Μόνικα Φρασόνη, στην οποία δίνω το λόγο τώρα. Μόνικα Φρασόνη, Φρασόνη ήταν και μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 5η και την 6η θητεία. Ήταν συμπρόεδρος με τον κ. Κομπέντη των Πρασίνων και της Φιλελεύθερης Συμμαχίας και όσον αφορά τα κόμματα, είναι συμπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος μαζί με τον Φιλίπ Λαμπέρ. Λοιπόν, Μόνικα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είμαι πολύ ικανοποιημένη που έχω τη δυνατότητα και την ευκαιρία να επιστρέψω σε αυτή την αίθουσα που επί 10 χρόνια ήταν η επιτροπή μου. Λοιπόν, πραγματικά είμαι πολύ ευχαριστημένη που είμαι εδώ ανάμεσά σας σήμερα το πρωί. Θα ήθελα εν ονόματι του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος και του συμπροέδρου μου, του Φιλίπ Λάμπερτς, που αναφέρατε. Οι πράσινοι έχουν αυτή τη συνήθεια που πιστεύουμε ότι είναι πολύ ε, καλή να έχουμε επικεφαλής δύο προέδρους για να υπογραμμίσουμε και να ενισχύσουμε ε, την ισότητα των φύλων και να μοιραζόμαστε και τις αρμοδιότητες και να εργαζόμαστε περισσότερο και καλύτερα. Εν ονόματι του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος έχω κάποιες παρατηρήσεις που εν μέρη ήδη αναφέρθηκαν από τους συναδέλφους που πήραν το λόγο πριν από μένα. Πρώτο στοιχείο αφορά το θέμα του νομικού καθεστώτος. Το νομικό καθεστώς είναι ένα θεμελιώδη στοιχείο όσον αφορά την ταυτότητα μιας ενώσεως, ενός κόμματος όπως είναι η δική μας περίπτωση. Το ότι εμείς δεν είμαστε ευρωπαϊκές ενώσεις, ευρωπαϊκά κόμματα αναγνωρισμένα ως τέτοια, μας στερεί από ένα θεμελιώδη στοιχείο ε, της δυνατότητας που μπορούμε να έχουμε να δράσουμε και τη ταυτότητά μα όσον αφορά του Ευρωπαίου πολίτε, έναντι των οποίων εμεί πάνω απ' όλα, πρώτα απ' όλα θέλουμε να μιλάμε ε, και για αυτού θέλουμε να κινούμεθα και να δρούμε. Λοιπόν, η κυρία Νέιτ είπε ότι δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα νομιμότητα όσον αφορά τα κόμματα, όμω το καθεστώ το νομικό δεν είναι ένα στοιχείο γραφειοκρατικού χαρακτήρα, είναι, συνταγματι... είναι βασικό στοιχείο, συστατικό στοιχείο τη ταυτότητά μα. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο εμεί σίγουρα και το προωθούμε κι εμεί άλλωστε, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ενωμένοι, διότι πιστεύω ότι είναι θεμελιώδε στοιχείο. Ε, κατανοώ και θα ήθελα επ' αυτού να διεξαχθεί μια συζήτηση ανοιχτή ε, με του φίλου μα και συναδέλφου των ε, Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν προβλήματα, διεξάγονται συζητήσει. Ήμουνα σε αυτό το σώμα και επί σειρά ετών παρακολούθησα το θέμα του ενιαίου καθεστώτος των βουλευτών, του ενιαίου καθεστώτος των βουλευτών Άρα γνωρίζω ότι υπάρχουν δυσκολίες. Όμως ε, πιστεύω ότι αυτές οι δυσκολίες που ουσιαστικά είναι γραφειοκρατικές θα πρέπει να ξεπεραστούν διότι στόχος πιστεύω ότι είναι ένας στόχος που δεν μας επιτρέπει να έχουμε μεταξύ πολιτικών κομμάτων και ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ανταγωνισμό ε, σε επίπεδο γραφειοκρατικό. Και πιστεύω και ελπίζω ότι από αυτή την πλευρά θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία που θα μας επιτρέψει να παρουσιάσουμε ένα νέο μέτωπο όσον αφορά τους άλλους θεσμούς για να πετύχουμε αυτό το νομικό καθεστώς, το νόμιμο καθεστώς. Θέλουμε επιμείνουμε και επί δύο σημαντικών στοιχείων που ίσω διεφάνισαν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. Δηλαδή, ο ρόλο που έχουν οι ενώσει ή οι ομάδε των νέων, youth organizations των κομμάτων και τα διάφορα ιδρύματα. Και τα δύο στοιχεία θα πρέπει να αναγνωριστούν περισσότερο διότι αποτελούν συστατικά στοιχεία τμήματα των δράσεων που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα ιδρύματα αυτά, οι ενώσεις, είναι κρίσιμο στοιχείο ε, διαμόρφωσης της σκέψης και ένας θεός ξέρει πόσο η διαμόρφωση της ευρωπαϊκής σκέψης ε, έχει, είναι λιματική σήμερα. Λοιπόν, η κοινή δουλειά της πολιτικής με τα πανεπιστήμια και γενικά με τα ιδρύματα και προφανώς και με την συμμετοχή των νέων Όλα αυτά θα πρέπει να αξιοποιηθούν από την προσπάθειά μας και εμείς απράσινοι, πιστεύουμε ότι αυτά τα στοιχεία είναι πραγματικά σημαντικά. Συμφωνώ με το θέμα της ύπαρξης τουλάχιστον ενός ευρωβουλευτού, αλλά όσον αφορά τη χρηματοδότηση για αυτό το θέμα, για την χρηματοδότηση, όχι την αναγνώριση. Πιστεύουμε ότι όσον αφορά την αναγνώριση, αξίζει πολύ περισσότερο η αξία, ε, η παρουσία σε πολλές χώρες σε σχέση με την παρουσία στο Ευρωπαϊκό κυρίως αν μιλάμε για ένα και μόνο βουλευτή που προέρχεται από ένα κάτος μέλος, από τα κάτι μέλη. Πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο, πραγματικό περιθώριο, χώρος και ελπίζω αυτό το Κοινοβούλιο και είμαι σίγουρη ότι το Κοινοβούλιο το εκτιμά αυτό. Υπάρχει δυνατότητα λοιπόν υποστήριξης, κινητοποίησης, συμμετοχής των ευρωπαϊκών κομμάτων στις εκστρατείες, όχι μόνο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και εκστρατείες σημαντικές διαφόρων ευρωπαϊκών θεμάτων. Έχω να σας δώσω δύο παραδείγματα που θεωρώ σημαντικά. Ένα παράδειγμα είναι αυτό της συγκεκριμένης εφαρμογής της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Έγινε συζήτηση όσον αφορά την ελευθεροτυπία, δεν θέλω να επισέλθω επί της του θέματος, αλλά είναι προφανές ότι το Ευρωπαϊκό Κόμμα, τα ευρωπαϊκά κόμματα μπορούν να καταφέρουν πραγματικά να, να δημιουργήσουν συζητήσεις επικοινών θεμάτων που μπορούν να καλλιεργήσουν και να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν τις συζητήσεις που διεξάγονται εδώ και από τη φύση τους αυτές οι συζητήσεις είναι ευρωπαϊκής φύσεως. Πιστεύω λοιπόν ότι σίγουρα το νομικό καθεστώς ή τα θέματα της χρηματοδότησης που ήδη ανέφεραν οι συνάδελφοί μου και επέμειναν επί κάποιων πτυχών και εγώ βεβαίως συμφωνώ με αυτά είναι όλα αυτά στοιχεία που εξυπηρετούν, χρησιμεύουν στην αύξηση της δημοκρατίας στην Ήπειρό μας και να βελτιώσουν τη συμμετοχή των πολιτών. Να μην είναι κάτι εικονικό και θεωρητικό, αλλά είναι κάτι συγκεκριμένο όσον αφορά τα διάφορα συγκεκριμένα θέματα που οι πολίτες μας αντιμετωπίζουν σε εθνικό και προφανώς περιφερειακό επίπεδο. Και από αυτή την έποψη, λοιπόν, η συμμετοχή σε εκστρατείε και σε εθνικές και στα δημοψηφίσματα σίγουρα θα πρέπει να το μπορούμε να το εγγυηθούμε και στα ευρωπαϊκά κόμματα. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ λέει Πρόεδρος και τώρα να δώσω το λόγο στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αριστεράς που εισέλθει στο συνέδριο τη 5 Δεκεμβρίου του 2010, είναι πρόσφατο το καθήκον που ανέλαβε, στον Πιέρ Λοράν, ο οποίο είναι δημοσιογράφος, ε, γάλλο, ε, πρώην διευθυντή της Humanité, γενικός γραμματέας του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος και επαναλαμβάνω από τον περασμένο Δεκέμβριο είναι και πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Αριστερά. Έχετε το λόγο λοιπόν. Σα ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν φυσικά τον πρόεδρο Κασίνη και την κυρία Γιαννάκου για τη διοργάνωση αυτής της δημόσια ακρόσης. Το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς ιδρύθηκε πριν από έξι χρόνια και μόλις τον προηγούμενο Δεκέμβριο ανέλαβα εγώ την Προεδρία στο τέταρτο συνέδριο του κόμματος που αποτέλεσε μια σημαντική φάση στη ζωή του κόμματό μα και θέλουμε να προωθήσουμε τη δραστηριότητα του κόμματο Ευρωπαϊκή Αριστερά για πολλού και διάφορου λόγου. Καταρχήν, πιστεύω ότι ο ρόλο των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων είναι πολύ σημαντικό για το θέμα τη ευρωπαϊκή δημοκρατία, γιατί το θέμα αυτό ήταν, είναι και θα είναι κεφαλαιόδου σημασία γιατί η κρίση πραγματικά διέλυσε όλες τις προκαταλήψεις και τις διαμορφωμένες ιδέες. Θα πρέπει να επινοήσουμε καινοτόμες ιδέες στην Ευρώπη και χρειαζόμαστε ένα σωστό πλαίσιο για την συμμετοχή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα αυτά. Και αυτό θα αποτελέσει το μέλλον κέριο ζήτημα, γιατί χωρίς μια, ένα στέρεο ε, δημοκρατικό θεμέλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κίνδυνος κλειδονισμού είναι ακόμα μεγαλύτερος. Κατά τη γνώμη μας, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα διαδραματίσουν εξέχοντα ρόλο στη διαδικασία αυτή. Ποια είναι η αντίληψή μας τώρα για την εξέλιξη αυτών των κομμάτων. Θα πρέπει καταρχήν να μην απομακρύνουμε αυτά τα κόμματα από τους πολίτες, να μην στραφούμε μόνο στην ηγεσία τους, θα πρέπει να έχουμε ευρωπαϊκά κόμματα που θα συνδέονται στενά με τους πολίτες και θα αντανακλούν πραγματικά τη γνώμη τους και θα τους αντιπροσωπεύουν. Θα δίνουν ουσιαστικά φωνή και δυνατότητα επιρροής και επέμβαση στον Ευρωπαίο πολίτη. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα πρέπει να παραμείνουν ε, ως ε, συνασπισμοί διαφόρων πολιτικών κομμάτων και τα μέλη τους ε, και οι Ευρωπαίοι πολίτες θα διαδραματίζουν στην δομή αυτών των κομμάτων ενεργό ρόλο. Ο πρωταρχικός στόχος των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων θα πρέπει στις σημερινές συνθήκες να είναι να αισθανθούν οι πολίτες ότι έχουν ε, τον έλεγχο αυτών των κομμάτων και ότι συμμετέχουν στην επιλογή των ευρωπαϊκών προκλήσεων και θεμάτων. Σε ό,τι αφορά την κύρωση της συνθήκης, για παράδειγμα. Δεν μιλώ για το αποτέλεσμα, αλλά είχαμε ήδη την εμπειρία μια συζήτηση και ενό δημοψηφίσματο για την Ευρωπαϊκή Συνταγματική Συνθήκη στη Γαλλία. Θα ήθελα να σας το υπενθυμίσω γιατί είναι σημαντικό να θυμηθούμε αυτά που είχαμε, είχε πει τότε ο ζαν κλοντ Γιούνκερ τις παραμονές του δημοψηφίσματο. Είπε ότι η προοπτική του δημοψηφίσματος ε, ξεκίνησε στη Γαλλία μια πολύ σημαντική συζήτηση, πολύ ποιοτική, γιατί η Ευρώπη δεν είναι πια προνόμιο των ελίτ, αλλά στη συζήτηση αυτή συμμετέχει και ο πολίτης, συμμετέχει και ο λαός, κάτι που δείχνει ότι ο λαός δεν αδιαφορεί για ένα θέμα όπως είναι το δημοψήφισμα, αλλά παθιάζεται όλο και περισσότερο γι' αυτό. Νομίζω ότι αυτό χρειαζόμαστε στην Ευρώπη όλο και περισσότερο, την ενεργό ανάμειξη του πολίτη και η εμβάθυνση του πολιτικού βίου των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων είναι κέριο ζήτημα και αφιερώσαμε πολλές, πολλές ώρες στο θέμα αυτό και στο τελευταίο μας συνέδριο και πολύ έργο. Θα πρέπει πραγματικά να συνδέσουμε τους πολίτες, ε, τα μέλη του κόμματος με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Είμαστε υπέρ μάλλον ενός νομικού πλαισίου που θα ενισχύει το ρόλο αυτών των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, όπως ανέφεραν και οι προλαλήσαντε, στο μέτρο που το νομικό αυτό καθεστώ θα εμπνέεται από τις καλύτερε δημοκρατικές παραδόσεις της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Θα πρέπει να εμβαθύνουμε λοιπόν ε, στη συζήτηση των συγκεκριμένων διατάξεων και ε, στον αντίκτυπό Σε αντίθεση με τους προλαλήσαντες, θα ήθελα να πω ότι η προοπτική ενός διακρατικού καταλόγου υποψήφιων ή επιλογή ευρωβουλευτών στα πλαίσια μιας ενιαίας εκλογικής, πανευρωπαϊκής εκλογικής περιφέρειας με ενιαίο κατάλογο ίσως δημιουργήσει προβλήματα απομάκρυσης των Ευρωπαίων πολιτών ε, σε αντίθεση με το στόχο μας που είναι η προσέγγιση. Δεν θα πρέπει να παρεκτραπούμε σε μια προσωποποίηση της ε, προεκλογικής εκστρατείας έχοντας κάποιες βεντέτες ε, στον κατάλογο. Θα πρέπει να ε, ενεργήσουμε υπέρ του πλουραλισμού και της προσέγγισης Ευρώπης προς τους πολίτες. Η θα διευρύνουμε το χάσμα αντί να το γεφυρώσουμε μεταξύ πολιτών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε μας βρίσκει σύμφωνος η άρση του ορίου των δωρεών σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις, οι επιδοτήσεις σήμερα είναι μάλλον πιο ευνοϊκέ για τα μικρά κόμματα όπως είναι το δικό μας, αλλά θα προτιμούσαμε να μείνουμε στις ε, σημερινές ε, αναλογίες 15%-85%. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, είμαστε υπέρ δύο εξελίξεων για να μπορέσουν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να είναι πιο δραστήρια στις εκλογικές εκστρατείες, προεκλογικές εκστρατείες, έχοντας αφενός τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που συνήθως είναι καρπός συνεργασίας μεταξύ ενός δύο περισσότερων κομμάτων μελών. Αυτή η συνεργασία θα πρέπει να προωθηθεί και να ενθαρρυνθεί και τα κόμματα μέλη που οργανώνουν τέτοιες πρωτοβουλίες για τα σημαντικά πολιτικά ζητήματα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν επιδότηση για τις πρωτοβουλίες τους, γιατί πραγματικά ενισχύουν την ε, πολιτική συζήτηση στην κοινή γνώμη. Φυσικά η προεκλογική εξαιρετή για τις ευρωεκλογές είναι πολύ σημαντική, γιατί η αποχή από τις εκλογές, από τις ευρωεκλογές ε, μας ενισχύει όλους, το μεγάλο ποσοστό αποχής. Θα πρέπει να αποκαταστήσουμε την ε, σημαντική παρουσία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δημόσια συζήτηση. Δεν είμαστε υπέρ της άρσης του, της χρηματοδότησης για την Ευρωπαϊκή Προεκλογική Εξηλατεία. Σας ευχαριστώ κύριε Λοράν. Προτείνω σε αυτή τη φάση αφού ακούσαμε πέντε από τις προσωπικότητές μας, από τις εννέα που συμμετέχουν στις εργασίες μας, να να κάνουμε να ακουστούν παρεμβάσεις, ερωτήσεις σύντομα από πλευράς μελών της Επιτροπής σε σχέση με την παρέμβαση των πέντε προσωπικότητων που ήδη μίλησαν. Και μετά μπορούμε να συνεχίσουμε μέσω παρεμβάσεων του κυρίου Ντεφούρτ, Κάτς, Κοτσιλόβο και Βανβίκ. Θέλετε να το κάνουμε έτσι. Αν κάποιος θέλει να πάρει το λόγο βέβαια. Θέλετε να πείτε κάτι ίσως. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα ε, τα στελέχη και τους υψηλόβαθμους των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων που προσήλθαν εδώ σήμερα για να εξετάσουμε επευκαιρία της χρηματοδότησης των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων του τρόπου χρήσης αυτών των χρημάτων που αποτυπώνονται στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα και ένα μεγάλο έλλειμμα το οποίο είναι καθαρά πολιτικό έλλειμμα είναι το πολιτικό έλλειμμα του να υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση με νομική προσωπικότητα και τα ευρωπαϊκά κόμματα να στερούνται νομικής προσωπικότητας ή να είναι μη κυβερνητικέ οργανώσεις διεθνούς χαρακτήρα στις Βρυξέλλες ή και αν θέλετε εάν η επιθυμία τους είναι να είναι εγκατεστημένα σε κάποιες άλλες χώρες της Ένωσης να έχουν την έδρα τους να μπορούν να το κάνουν υπό ίσους όρους. Εγώ θέλω να εκφράσω την ε, χαρά μου διότι όλοι όσοι μίλησαν ξεκαθάρισαν ότι αυτό είναι αναγκαιότητα ότι είναι κάτι που λείπει και ότι μας χρειάζεται πολιτική, νομική ε, και φορολογική ε, αρχή επί της οποίας θα βασίζονται τα ευρωπαϊκά κόμματα. Δεν έχω να κάνω ερωτήσεις κύριε Πρόεδρε, απλώς ήθελα να εκφράσω κι εγώ τη συμφωνία μου με όσα ελέγχθησαν λεπτομέρειες για τη χρηματοδότηση πόσο πάνω θα είναι ή πόσο κάτω κτλ. Αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε και πάλι και να τα δούμε. Σημασία έχει ότι αρχίζει να δίνεται το μήνυμα ότι έχει φτάσει ο χρόνος να υπάρξει πραγματικά αυτή η σοβαρή πολιτική κίνηση και αν θέλουμε να ενισχύσουμε και την παρουσία των πολιτών μας και στις ευρωεκλογέ, δηλαδή να έρχονται να ψηφίσουν γιατί πια το ποσοστό αποχής αυξάνεται συνεχώς αλλά και να ενδιαφερθούν για τα ευρωπαϊκά πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ντάφελη να πει κάτι τώρα. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όσους μίλησαν εξ των πολιτικών κομμάτων και με την ιδιότητά μου ως ε, συγητής για τη μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας του Κοινοβουλίου. Ελπίζω να υπάρξει μια μεταρρύθμιση μέχρι το 2014. Βασικό μέρος των προτάσεων που έχουμε είναι, όπως ξέρετε, να δημιουργήσουμε ένα πανευρωπαϊκό εκλογικό σώμα, να εκλέξουμε άλλους 25 ευρωβουλευτές από διεθνείς υπερεθνικές λίστες και στόχος όλων αυτών και βασικός στόχος πρότασης είναι να σφυριλατηθεί να σφυριλατηθούν ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα γιατί είναι καλές οι αλλαγές νομικές και απαραίτητες, πρέπει να γίνουν, αλλά αυτό το οποίο θα μεταμορφώσει αυτά τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή, όσο σεβαστά και αν είναι, αλλά με κάθε σεβασμό ακόμη πρωτόγωνα, αυτό το οποίο λοιπόν θα τα μεταμορφώσει σε πραγματικά πολιτικά κόμματα, οργανισμούς που θα κάνουν εκστρατείες, είναι να επιβληθεί το καθήκον να βρουν, να επιλέξουν και να κατατάξουν υποψηφίους από το Ευρωπαϊκό, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να δημιουργηθούν δηλαδή λίστες, να κάνουμε εκστρατείες για ιδέες, για πολιτικές, για έδρες και για ψήφους. Και νομίζω πως η πρόταση που βρίσκεται ενώπιον του Κοινοβουλίου είναι επαρκής για να μεταμορφώσει την ε, κομματική κατάσταση στο ομοσπονδιακό επίπεδο. Να είμαστε ειλικρινεί για το τι προσπαθούμε να επιτύχουμε. Εγώ θεωρώ την δημιουργία ομοσπονδιακών πολιτικών κομμάτων ως βασικό μέρος ε, της μεταεθνικής δημοκρατίας. Και ως μέρος του μεταρρυθμιστικού πακέτου. Σημαντικό είναι να επιμείνουμε πως καθώς ενηλικιώνονται τα ομοσπονδιακά πολιτικά κόμματα μπορούν να διασφαλίσουν πρώτης τάξεως εσωκομματική δημοκρατία και όσον αφορά τις εσωτερικές τους διαδικασίες για την επιλογή υποψηφίων αλλά βεβαίως και όσον αφορά την οικονομική διαφάνεια και λογοδοσία. Ένα τρίτο στοιχείο. Και θα ήμουν ευγνώμων ε, εάν θα μπορούσα να αναφερθώ σε αυτό προσωπή των πολιτικών κομμάτων. Είναι η δημιουργία ενός τμήματος για να μπορούν να γίνουν μέλη απευθείας οι πολίτες. Δεν αρκεί τα πολιτικά κόμματα να συναποτελούνται από εθνικά πολιτικά κόμματα. Δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε τα εθνικά κόμματα. Ε, ζητάμε όμως να τα συμπληρώσουμε με κάτι το διακριτό, ρητό με την άμεση εμπλοκή των πολιτών στην μεταεθνική δημοκρατία. Και θα αποτελέσει αυτό βασικό μέρος της μεταρρύθμισης των πολιτικών κομμάτων που θα προκύψει από την υπερεθνική λίστα να έχουν όλα τα κόμματα ένα αποτελεσματικό μηχανισμό για την εγγραφή μελών άμεσα που θα πληρώνουν συνδρομή στο Ομοσπονδιακό Πολιτικό Κόμμα ως κάτι το διακριτό από τους πολίτες που εμπλέκονται στα εθνικά κόμματα όπως θα επιλέξουν κάποιοι να κάνουν. Αλλά κάποιοι άλλοι θα επιλέξουν να μην ε, γίνουν μέλη εθνικού πολιτικού κόμματος. Κάποιοι θα επιλέξουν να εγγραφούν απευθείας στο Ομοσπονδιακό Κόμμα. Οπότε θα ήθελα να ακούσω από τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων ε, που θα μιλήσουν εάν θεωρούν κάτι τέτοιο ε, ως κάτι το εφικτό στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Προτείνω σε αυτή τη φάση να μιλήσουν οι συνάδελφοι Χέφνερ και Γκρότ που ζήτησαν να παρέμβουν, αλλά άλλοι συνάδελφοι ας μιλήσουν στο τέλος μετά τις επόμενες παρεμβάσεις από πλευρά πολιτικών κομμάτων, διότι έχουμε να ακούσουμε τέσσερα άτομα. Λοιπόν, και ο Χέφνερ πρώτα και παρακαλώ Εστέλα Κονικός. Ich kann das allerdings gerne auch... Κοιτάξτε, μπορώ να τοποθετηθώ και στο δεύτερο γύρο, αν θέλετε, όταν ακούσουμε, όταν τους έχουμε ακούσει όλους. Al presidente στον πρόεδρο Ερικ Ντεφούρ, που είναι πρόεδρος του Λαϊκού κινήματο, πρόεδρος της Φιλελεύθερης Ευρωπαϊκής Συμμαχίας, ήταν πρόεδρος του ε, φλαμανδικού λαϊκού κινήματος και καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τώρα βρισκόμαι μεταξύ σας, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. ελπίζω να μην ε, υπάρχει κανένα πρόβλημα στο να παρέμβω μετά τους ε, συναδέλφους. Λοιπόν, τώρα βρίσκομαι... Ήμουν. Εξελέγει, με συγχωρείτε, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ελευθερής Συμμαχίας το Μάρτιο του 2010 στο συνέδριο στην ε, Βενετία διάδοχος κυρίας Νέλη Μάση η οποία ήταν επί σειρά ετών Ευρωβουλευτής και το κόμμα του οποίου προεδρεύω αυτή τη στιγμή δεν είναι από τα μεγάλα κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά είναι οπωσδήποτε ένα ολοκληρωμένο κόμμα. Αν θέλετε, συστάθηκε το 1981 και ορτάζουμε βεβαίως φέτος τα 30 έτη μας και ως πραγματική, πραγματικό και φιλοευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα μπορώ να σας πω πως έχουμε έξι κράτη, έξι ε, μέλη από πέντε κράτη-μέλη και έχουμε 7 ε, ευρωβουλευτές, 8, 8 κόμματα με εθνικούς βουλευτές και εκπροσώπους επίσης σε περιφερειακά κοινοβούλια. Και βεβαίω αν εφαρμοστούν αυτά τα οποία ακούμε σήμερα θα ενταχθούμε οπωσδήποτε και θα ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία Άκουσα με ιδιαίτερη ικανοποίηση τους προλαλήσαντε και θα μου επιτρέψετε λίγο σοβενισμό και με ιδιαίτερη ικανοποίηση τον συμπατριώτη μου, τον κύριο Βίλφρυντ Μαρτέν, αλλά και την κυρία Μόνικα Φρασόνη και η παρατήρησή της όσον αφορά τι νεολαίε των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Νομίζω πως ε, οι σκέψει ε, της κυρία Φρασόνη εκεί πέρα ήταν πάρα πολύ σημαντικέ, ειδικά από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία. και βεβαίως από πλευράς νεολαίας αλλά και παρουσία στην ευρωπαϊκή κοινωνία αν δούμε τώρα τις προτάσεις ε, που υπάρχουν μέσα σε αυτή την έκθεση εμείς ως Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία έχουμε κάποιες σκέψεις ε, όχι ύψο φακτο επικριτικές αλλά κάπως ε, θα έλεγα επιφυλακτικές. Και θα ήθελα λοιπόν να δώσω τον λόγο στον διευθυντή μας που κάθεται στα αριστερά μου για να εκφράσει κάποιες από αυτές τις σκέψεις. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Συγητά, θα ήθελα να αναφέρω κάποιες σκέψεις που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, τον εκδημοκρατισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια τη μεταρρύθμιση της συζήτησης που γίνεται των θεσμικών οργάνων. Θεωρώ σημαντικό να πω πως στηρίζουμε την πρόταση για τα κριτήρια αναγνώρισης των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και για τον καλύτερο ορισμό τους. Στηρίζουμε δηλαδή το ότι κατά κανόνα θα αναγράφεται πως πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας ευρωβουλευτής ε, για να στηρίζει αυτό το Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα για να υπάρξει μια αναγνώριση και πράγματι αυτό συμβαίνει και η έρευνα έχει δείξει πως ε, αυτή η έρευνα την οποία ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας του Κοινοβουλίου και πράγματι αρκεί ε, σε μεγάλο αριθμό κρατών μελών να υπάρχει ένας ευρωβουλευτής για να υπάρχει αυτή η ε, αναγνώριση. Πράγματι είναι σημαντικό να γραφτεί αυτός ο κανόνες, αλλά θα πρέπει να πούμε πως δεν μπορεί να είναι αυτό το πρώτο βήμα για ε, να έχουμε περισσότερους ευρωβουλευτές για να έχουμε ένα κατόφλι αν θέλετε για την αναγνώριση. Νομίζουμε καλό θα είναι να έχουμε την ε, χρηματοδότηση. Εντάξει, η χρηματοδότηση το αντιλαμβανόμαστε ότι θα είναι κατά ένα 85% της 100 καταναλογία με το μέγεθος, ε, όπως ακριβώς συμβαίνει και στα κρατημέλη. Επίσης στηρίζουμε το ότι τα κόμματα δεν θα μπορούν να αναγνωριστούν ως ευρωπαϊκά ε, πολιτικά κόμματα βασισμένα μόνο σε άτομα. Θα πρέπει να είναι διεθνείς οργανισμοί που θα έχουν ως μέλη τα κόμματα. Τρίτο και σημαντικό, κύριε Πρόεδρε, βρίσκουμε πάρα πολύ σημαντικό να εκπροσωπείτε το περιφερειακό επίπεδο στα κριτήρια αναγνώρισης. Αυτό είναι σημαντικό για τον εκδημοκρατισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι πλήρως στο πνεύμα της Συνθήκης Λισαβόνας. Και τέλος, η ποικιλία ποικιλομορφία της συζήτησης ε, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Θεωρώ πως ε, οι σημερινές ε, συζητήσεις αντικατοπτρίζουν μια καλή ισορροπία για να μην έχουμε κατακαιρματισμό της ευρωπαϊκής συζήτησης με πάρα πολλούς εταίρους, αλλά να εγγυώνεται βεβαίως πλήρως και την ποικιλομορφία της συζήτησης. Οπότε είναι οι σημερινές προτάσεις ε, αρκετά ε, ισορροπημένες, αλλά αν υπάρχει κάποια αλλαγή στο μέλλον θέλουμε να το έχετε αυτό κατά νου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τους δύο εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμμαχίας και τώρα ο κύριος Άσπερ Κάτς που είναι διευθυντής τη Συμμαχία των Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, των Ευρωπαίων Συντηρητικών Μεταρρυθμιστών. Είχε το λόγο. Ε, thank you very much, Chairman. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη, διότι ούτε ο Πρόεδρος μου, ο Γιάν Σάρντελ, ούτε ο Γενικός Γραμματέας Νταν Χάναν μπόρεσαν να παραστούν σήμερα. Το ACR δημιουργήθηκε μόλις πριν από ένα χρόνο, το κόμμα μας, Οπότε είμαστε το... ο Βενιαμίν της οικογένειας, ο νέος. Γι' αυτό θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Και έχω δύο παρατηρήσεις μόνο. Μία επί της αρχής και μία πρακτικής μορφής. Τα εθνικά κόμματα στο προβλεπόμενο μέλλον θα έχουν την πολιτική νομιμότητα αν θεσπίζουν νομοθεσία. Οπότε βελτιώνεται ελάχιστα η δημοκρατική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αν επιτραπούν στα πολιτικά, ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να ε, προσπαθήσουν να κάνουν προεκλογική στρατεία για αυτά κάθε αυτά. Δεύτερον, όσον αφορά το ευρωπαϊκό επίπεδο, το πώς θα κυβερνώνται αυτά τα πολιτικά κόμματα, για κάποιον που είναι καινούριο, είναι ασαφής η κατάσταση σε πολλές περιπτώσεις και δύσκολο να ε, ερμηνευθούν για νέους φορείς. Είναι δυσ, δυσνόητοι οι κανονισμοί. Άρα χρειάζεται βελτίωση της διαφάνειας και της αφήνειας των κανονισμών, των κανόνων, κυρίως όσον αφορά το ποια θα είναι η πρακτική που καθιερώνεται. Από τη στιγμή που καθιερώνεται μια πρακτική, δύσκολο να ανακαλύψει κανείς ποιες είναι αυτές οι πρακτικές. πολλή ενέργεια λοιπόν πρέπει να διατεθεί προς διευκρίνηση των ζητημάτων αυτών. Όμως καταλαβαίνω γιατί είναι πρακτικόν οι παλιοί οργανισμοί να έχουν αυτή τη δομή και εμείς ανεφέ το χρόνο είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνήσουμε με αυτή την προσέγγιση. Και όσο θα μαθαίνουμε και θα προοδεύουμε, είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε περισσότερα σχόλια και θα τα υποβάλουμε γραπτός. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον κύριο Κοτσιλόβο που υπήρξε μέλος του κοινοβουλίου μας και ήταν και αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ευρωπαϊκού και είναι γενικός γραμματεύς του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ εν ονόματι του κόμματος που εκπροσωπώ σας ευχαριστώ εσάς, τα μέλη της Επιτροπής και προφανώς την κυρία Γιαννάκου που ανέλαβε αυτή την έκθεση και μοιραζόμαστε, συμμεριζόμαστε τις βασικές γραμμές. Διευκολύνεται το έργο μου, διότι ήδη άκουσα παρεμβάσεις με τις οποίες συμφωνώ σχεδόν απόλυτα. Υπήρξε και προηγούμενο μια κοινή επιστολής που υπεγράφει από όλα τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και απεστάλλει στο Γενικό Γραμματέα στα πλαίσια της ετήσιας διαδικασίας ε, για την έκθεση για τη χρηματοδότηση των κομμάτων. και θεωρείται δεδομένο το περιεχόμενο της επιστολής και συγκλίνουμε και επί των διαφορών προτάσεων. Θεωρώ εξάλλου σαφές, διαφάνηκε από τις πρώτες παρεμβάσεις και από αυτές που ακολούθησαν και από αυτά που υπόθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής ότι η σημερινή ακρόαση ξεπερνά έναν απλό προβληματισμό όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού η χρηματοδότηση των κομμάτων για τη διαδικασία, τα προβλήματα που μπορεί να ξεπεραστούν, αλλά θέλουμε να δούμε μέσω της αναγνωρίσεως του ρόλου των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων μπορούμε να ολοκληρώσουμε ένα οικοδόμημα κοινοτικής ηθαγένειας, ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Κάτι που παραμένει στόχος και όραμα πολιτικό της πλειοψηφίας των κομμάτων. Και πρέπει να υπογραμμίσω κι εγώ όπως και άλλοι ότι είναι κατεπήγον να κατακτήσουμε ένα κοινό καθεστώς ευρωπαϊκό. Ένα νομικό πλαίσιο αναφοράς με άλλα λόγια για ιδρύματα και κόμματα. που μπορεί να συνδέεται με το νόμο και το πλαίσιο της Ένωσης. Ακούστε ικανά απόψεις για αυτό το στόχο, προσεγγίσεις, σκέψεις. Θα ήταν απλό να δοθούν και κάποιες λύσεις και συγκεκριμένο πρόβλημα, πιστεύω που εντοπίστηκε. Τη δυνατότητα το προσωπικό των κομμάτων και των ιδρυμάτων να μπορεί να ενταχθεί σε ένα φορολογικό καθεστώς που ήδη έχει οθετηθεί όσον αφορά υπαλλήλου των κοινοτικών οργάνων και άλλων και του υπόλοιπου προσωπικού. Πρέπει να υπάρξει εγγύηση ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, την ευρωπαϊκή για τα κόμματα, πρέπει να συνδέεται με την παρουσία τουλάχιστον ενός Ευρωπαίου βουλευτού και συμφωνώ με τις εκφραστήσεις απόψεις που αποσυνδέουν αυτό το στοιχείο από τη διαδικασία και το αποτέλεσμα της αναγνωρίσεως του Ευρωπαϊκού Κόμματος. Μπορεί να υπάρχει αναγνώριση μέσω άλλων στοιχείων που ήδη αναφέρθηκαν για τη χρηματοδότηση. Πέρα από τα... Δηλαδή, διαχωριστή η χρηματοδότηση λοιπόν από την ελάχιστη κοινοβουλευτική αντιπροσώπευση που απαιτείται για τη χρηματοδότηση. Εν ώψη κοινού ρυθμιστικού πλαισίου. la possibilità di adesione diretta. Λοιπόν και την δυνατότητα άμεση συμμετοχή ε, απομονωμένων, μεμονωμένων βουλευτών ή πολιτών Ακούστηκαν διάφορες θέσει επ' αυτού. Και από την παρέμβαση του κυρίου Νταφ ακούσαμε κάποια στοιχεία. Ας αφήσουμε εκτός την κοιλωτίνα που θα μπορούσε να θέσει τροχοπέδι στην άμεση συμμετοχή των πολιτών σε επίπεδο εκπροσώπησης δευτέρου βαθμού, δηλαδή εκπροσώπηση στις διάφορες χώρες ενός κόμματος που προσχωρεί σε Ευρωπαϊκό Κόμμα. Χρειάζεται διαφανής κάλυψης συμμετοχής των πολιτών άμεσης και των βουλευτών. Αυτό αν γίνει είναι ένα στοιχείο που υποστηρίζει το ρόλο και το σκοπό των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Στην προσπάθεια οικοδόμησης της κοινής ηθαγένειας. Δεν πρέπει να υπάρχει διπλή συμμετοχή Προφανώς δεν θα πρέπει ένας που είναι σε ένα κόμμα να προσχωρήσει μετά σε άλλο ευρωπαϊκό κόμμα. Ή για βουλευτές που εκλέγονται από τη λίστα και που ανήκουν σε κόμμα να προσχωρήσουν σε άλλα ευρωπαϊκά κόμματα. Λοιπόν, η διπλή εγγραφή θα πρέπει να αποφεύγεται. Θέλω να υπογραμμίσω τη δυνατότητα άμεσης συμμετοχής σε εκστατήσια δημοψηφίσματα και πιο αποφασιστικό ρόλο στις πολιτικές εκστρατείες ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Όσο αφορά τη διαδικασία για τη χρηματοδότηση κλπ. Υπάρχουν ρυθμίσεις που μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό για τα ιδρύματα να μην υπάρχει όμως εκεί το εμπόδιο όσον αφορά την βοήθεια μέσω ιδίων πόρων για τη χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειάζεται και απλούστευση των διαδικασιών. Γι' αυτό εμπεριέχεται στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα ε, κάτι συγκεκριμένο. Να αποφύγουμε δημιουργία εμποδίων διότι, λόγω περίπλοκων ε, διαδικασιών χρειάζεται να επικρατήσει διαφάνεια. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Κατά τα λοιπά, για λεπτομέρειες, μπορείτε να δείτε και την επιστολή που απέστελαν τα πολιτικά κόμματα στο Γενικό Γραμματέα. Ευχαριστώ κύριε Κοτσιλόβο. Τελευταία παρέμβαση τώρα, όσον αφορά τα κόμματα. Ο κύριος Δίκ Βαντίκ, που είναι ε, υπεύθυνο τα οικονομικά θέματα για του, του χριστιανικού Ευρωπαϊκού Κόμματο. Ταμεία του κόμματο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη τη Επιτροπή, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να σχολιάσω την έκθεση του Γενικού Γραμματέα για τη χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων. Μα ικανοποιεί γενικώ η έκθεση, βέβαια μπορούν να γίνουν κάποιε βελτιώσει στι διαδικασίε. Επίση μα. Ε, βρίσκει η δήλωση ότι στόχος της ρυθμής αυτής είναι να φτάσει όσο το δυνατό περισσότερους δικαιούχους η χρηματοδότηση. Θα ήθελα να περιοριστώ στο, σε ένα ζήτημα της ε, σελίδας 27 της έκθεσης που μιλάει για τις υποχρεωτικές διαστάσεις ενός Ευρωπαϊκού Πολιτικού Κόμματος προκειμένου να είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση. Εμείς Μόνο από πέρυσι έχουμε κερδίσει αυτό το χαρακτηρισμό του Ευρωπαϊκού Πολιτικού Κόμματο, οπότε μπορούμε να καταθέσουμε την εμπειρία μα. Η εμπειρία μα είναι ότι ισχύουν κανονισμό, ιδιαίτερα το άρθρο 3.1β, που αναφέρει ότι ένα πολιτικό κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να πληρεί την προπόθεση ότι θα πρέπει να εκπροσωπείται σε ένα τέταρτο των μελών, από, να εκπροσωπείται από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή από εθνικού βουλευτέ ή σε τοπικέ βουλέ. Ο κανονισμό αυτό είναι ήδη αρκετά περιοριστικός για ένα κίνημα όπως είμαστε εμείς, το Ευρωπαϊκό Χριστιανικό Κίνημα. Γιατί τέτοια κινήματα που έχουν ρίζες στην ευρωπαϊκή κοινωνία, όπως το δικό μας, και έχοντας υπόψη το στόχο ότι θα πρέπει να φτάσει η ρύθμιση όσο το δυνατό περισσότερους δικαιούχους, το κριτήριο αναγνώρισης δεν θα πρέπει να γίνει πιο αυστηρό. Ως εκ τούτου, το χριστιανικό κίνημα δεν μπορεί να ταχθεί υπέρ της ε, ακαδημαϊκής πρότασης πανεπιστημιακής των αιτιολογικών σκέψεων 85 και 86 που αν τεθούν σε εφαρμογή ουσιαστικά θα καταπνίξουν το δικό μας κίνημα και κατά πάσα πιθανότητα και κανένα άλλο κανένα δυο άλλα παρόμοια κινήματα με το δικό μας. Και η πρόταση να γίνει πιο αυστηρό το κριτήριο αναγνώριση, όπως προτείνει η έκθεση του Γενικού Γραμματέως, αντιβαίνει και στην ε, ε, επιθυμία των ε, υπαρχών των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Θα ήθελα να σας παραπέμψω στο παράρτημα 1 της έκθεσης που λέει ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θέλουν να προτείνουν αναθεώρηση του κριτηρίου αναγνώρισης και να προβλέπει ότι για την αναγνώριση και τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ευρωπαϊκό κόμμα θα πρέπει να εκπροσωπείται στην Ευρωβουλή, όπως ανέφεραν ε, η προλαλήσα της. Δηλαδή θα πρέπει τουλάχιστον να έχει έναν ευρωβουλευτή. Μία πιθανή τροπολογία του κριτηρίου αναγνώρισης, κατά τη γνώμη μας, δεν θα πρέπει να υπερβεί αυτή την πρόταση. Αυτά προς το παρόν κύριε Πρόεδρε. Θα σας στείλουμε και γραπτό στα σχόλιά μας και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε ερωτήσεις και να ακούσω τα σχόλιά σας. Grazie. Allora sono terminate eh, le relazioni. Le... Ευχαριστώ λοιπόν. Ακούσαμε τις απόψεις των πολιτικών κομμάτων που στην αίθουσα. Συνεχίζουμε τη συζήτηση με την παρέμβαση των μελών της Επιτροπής μας. Έφνερ και Γκρότ ζήτησαν το λόγο. Έχετε το λόγο. Κύριε Έφνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όσους μίλησαν για τις ουσιαστικές και χρήσιμες παρεμβάσεις. Μια παρατηρήση βεβαίως όλοι παίρνουν εξίσου αρά αυτά τα οποία λέγονται εδώ πέρα. Γι' αυτό και εγώ ε, ήθελα να μιλήσω αφού ε, ακουστούν όλοι οι συμμετέχοντες και όχι στο ενδιάμεσο. Τώρα, επί της ουσίας, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ και για την εξαιρετική προετοιμασία. Νομίζω μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα ένα μεγάλο βήμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ευρωπαϊκά κόμματα και όχι μόνο εθνικά. Παρά την καλή προετοιμασία, πιστεύω πως υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία πρέπει να συζητήσουμε εξαντλητικά. Πρώτα απ' όλα νομικές μορφές, προϋποθέσεις αναγνώρισης, χρηματοδότηση, προϋποθέσεις χρηματοδότησης, είναι επίσης ζητήματα εσωτερικής οργάνωσης των κομμάτων και το πώς παρεμβαίνει το εθνικό στο ευρωπαϊκό δίκαιο και αντιστρόφως. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στα βασικότερα αισθήματα και μετά να θέσω ερωτήσεις. Και κάτι άλλο ακόμα. Για μένα είναι αποφασιστικό το σε ποιο πνεύμα γίνονται όλα αυτά. Και βρισκόμαστε νομίζω σε ένα σταυροδρόμι γιατί εάν μιλάμε για την αναγνώριση ευρωπαϊκών κομμάτων, μιλάμε για βασικό συστατικό της δημοκρατίας. Η δημοκρατία χρειάζεται ανταγωνισμό και ο ανταγωνισμός χρειάζεται ως να δυνατόν πιο ανοιχτή πρόσβαση για περισσότερους. Και τι σημαίνει αυτό ότι θεωρώ πως κινδυνεύουμε να θεωρηθεί αυτό το οποίο κάνουμε ένα είδος κλειστής λέσχης για αυτούς που είναι ήδη μέσα και να κάνουμε πολύ δύσκολη την πρόσβαση σε αυτούς που θέλουν να μπουν. Δηλαδή, ε, επειδή είχα συνειδρήσει ένα κόμμα, τους πράσινους, και ξέρω από αυτή την ε, εμπειρία πως είναι σημαντικό οι νέες ιδέες να αναζητούν νέες μορφές και να παραμένει ο ανταγωνισμός πάντα και για εμάς που τώρα ανήκουμε στο κατεστημένο. Να μπορούμε ε, να αφήνουμε συνεχώς νέους να μπαίνουν. Οπότε υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία εδώ πέρα στο καθεστώς αυτό, στο σημείο όπου συνδέεται άρρηκτα το ζήτημα της αδειοδότησης με το ζήτημα της χρηματοδότησης. Γι' αυτό θα ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα. Μήπως είναι σημαντικότερο να ορίσουμε τρία διαφορετικά, τρεις διαφορετικές φάσεις νομικά. Πρώτα απ' όλα αδειοδότηση ως Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα υποευρωπαϊκή μορφή, όχι να γίνει βεβαίως ένας, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο, αλλά σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ειδικά αυτό όσον αφορά τα κόμματα, βεβαίω ισχύει και για ΜΚΟ κτλ. Πρώτον, η αδειοδότηση, όπου πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί, να επιτρέψουμε ευρύ ανταγωνισμό. Δεύτερον, ζήτημα συμμετοχή στι εκλογέ, όπου θεωρώ πως πρέπει να ισχύσουν πιο αυστηρές προϋποθέσεις, ε, ειδικά όσον αφορά τους επαρκείς, τον επαρκή αριθμό υποψηφίων και τρίτον και το ζήτημα της χρηματοδότησης που πρέπει να συνδεθεί με το ότι ένα κόμμα πρέπει να εργάζεται επαρκώς και η εργασία αυτή να στηρίζεται ε, επαρκώς από τον λαό. Ε, αυτά τα τρία στάδια έχουμε στην ε, Γερμανία και νομίζω πως σε μια τέτοια κατεύθυνση θα πρέπει να πάμε και εδώ πέρα όπως είπα για να μην θεωρηθούμε μια λέσχη αυτό που είναι ήδη μέσα και εμποδίζουν την πρόσβαση για τους υπόλοιπους. Οπότε δεν θα πρέπει να είναι μόνο η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προϋπόθεση, αλλά και συμμετοχή σε άλλο Εθνικό ή Περιφερειακό Κοινοβούλιο με νομοθετικές αρμοδιότητες. Και νομίζω εδώ πέρα κάτι σημαντικό είναι αυτό που ανέφερε νομίζω μόνο η Μόνικα Φρασόνη, δηλαδή η εσωτερική οργάνωση των κομμάτων. Α, με συγχωρείτε κι εσείς. Ε, να επιτραπεί δηλαδή ε, η αδειοδότηση των κομμάτων που είναι και στο εσωτερικό δημοκρατικά και ε, για τις αποφάσεις που λαμβάνουν και για την εκλογή σε αξιώματα και για την κατάρτιση των ληστών και ε, ο συνάδελφος ε, εδώ πέρα συγκατανεύει, ξέρετε πως έπρεπε να επαναληφθούν εκλογές στη Γερμανία γιατί ένα κόμμα που συμμετείχε σε αυτές τις εκλογές δεν είχε καταρτήσει τη λίστα με δημοκρατικές διαδικασίες αλλά κατόπιν απόφαση του Προεδρείου. Νομίζω λοιπόν πως χρειαζόμαστε ανάλογες προδιαγραφές στην Ευρώπη εάν είναι να έχουμε πανευρωπαϊκά κόμματα. Αυτά είναι τα σημαντικότερα σημεία που ήθελα να αναφέρω. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Γκρότε. Ευχαριστώ. Χαίρομαι για το ότι αφιερώνουμε τόσο πολύ χρόνο και χώρο για να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Είναι πακέτο ολόκληρο αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας για πολιτικά ιδρύματα. Επίσης πρέπει να μιλήσουμε αλλά ε, πρέπει να μιλήσουμε και για τους μη κυβερνητικού οργανισμούς που θα χρειάζονται ένα ανάλογο καθεστώς. Τέλος αυτό είναι μια άλλη συζήτηση αλλά πρέπει να το δούμε και αυτό και να κάνουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας. Όσον αφορά τη διαβάνεια, σήμερα άνοιξα μια μεγάλη γερμανική εφημερίδα η οποία έλεγε πως οι πολίτες στη χώρα μου δεν εμπιστεύονται ε, τόσο πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι την πολιτική, την επικοινωνία. Και αυτό πρέπει να το ακούσουμε. Δηλαδή αυτά τα οποία λέμε εμείς εδώ πέρα, αυτό το θέμα, να μεταφερθεί με διαφάνεια προς τα έξω και να υπάρξει μια λογική μετάδοση και επικοινωνία του γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάποιος αυτοσκοπός και αυτό το οποίο είπε ο κύριος Χέφνερ ε, είναι σημαντικό, δεν είναι να εξασφαλιστούν αυτοί που είμαστε, εμείς που είμαστε ήδη μέσα, αλλά να υπάρξει μια δημοκρατική βάση. Και αυτό είναι σημαντικό όσον αφορά τα οικονομικά. Νομίζω κύριος ε, Κοτσίλοβο μόνο ανέφερε, ε, δηλαδή τι θα γίνει με τους υπαλλήλου του κόμματος. Θα πρέπει να έχουν ένα καθεστώς όπως οι Ευρωπαίοι υπάλληλοι. Δεν το βλέπω. Εγώ δεν θεωρώ πως θα πρέπει να έχουν ένα ανάλογο καθεστώς. Γιατί δεν έχουν περάσει έναν διαγωνισμό ανάλογο. Είναι μια απόφαση ομόφωνη ε, του προεδρίου. Ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πως δεν θα πρέπει να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Να υπάρξει μια διάκριση. Γιατί δεν πρόκειται και για θεσμικό όργανο ούτως ή άλλως. Λοιπόν, επικοινωνία πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό πρέπει να το πούμε, σε, να συνοδεύσει ολόκληρη τη διαδικασία και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, το ανέφερε ο κ. μόλις. Εκεί πέρα πρέπει να διασφαλίσουμε πως θα υπάρξει μια δημοκρατική διαδικασία με κανόνες. Ε, είχαμε και την DAF. Είχαμε και την έκθεση DAF των σοσιαλιστών, αλλά βεβαίως έχουμε ένα τεράστιο πακέτο εδώ πέρα που πρέπει να ολοκληρώσουμε και πρέπει να δούμε πως ε, πρέπει να το διευρύνουμε σε ορισμένα σημεία, αλλά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε που έχουμε τον χρόνο να συζητήσουμε λογικά όλα αυτά τα ζητήματα. Νομίζω θα έχουμε ένα συναρπαστικό έτος μπροστά μας. Και τώρα δίνω το λόγο στον συνάδελφο Σόλτς. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γιαννάκου που ξεκινάει σήμερα νομίζω ένα μακροπρόθεσμο έργο που βεβαίω θα χαροποιήσει του φίλους της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Και κοιτάξτε, είναι ένα πολύ πολυπλοκό θέμα αυτό το οποίο βλέπουμε μπροστά μας και ακριβώς μετά από αυτά τα οποία είπαν οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ξέρετε κάποιοι από αυτούς ήταν και ευρωβουλευτές, θα έλεγα είμαστε φιλόδοξοι να μην κοιτάμε σε μικρή κλίμακα. Θα ήθελα να φέρω εγώ τρεις πτυχές που δεν έχω αναφέρθει όταν μιλάμε για την νομική υπόσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Το ζήτημα είναι πώς θα αναπτύξουμε ένα ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα κομμάτων. Δεν υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα αν είμαστε ειλικρινείς. Έχουμε εκπροσώπους των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων που βρίσκονται σε έναν κλειστό κύκλο του Κοινοβουλίου και έχουμε μετά κάτι το μιχλώδες, δηλαδή εξισώνονται τα πολιτικά κόμματα με την κοινοβουλευτική ομάδα. Αλλά αν θέλουμε να προχωρήσουμε σε ευρωπαϊκή δημοκρατία πρέπει να έχουμε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα τα οποία θα δρουν σε όλους τους τομείς στο ευρωπαϊκό και στο εθνικό επίπεδο υπό την έννοια κάποιου ο οποίος θα σχηματίζει την θέληση, θα επικοινωνεί όσον αφορά την πραγματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό το έχουμε συζητήσει και το τελευταίο έτος έτσι πλέον παρεμβαίνουμε στις ε, σχέσεις ισχύω μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και πρέπει να δούμε πώς θα είναι αυτές οι σχέσεις μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων στο μέλλον ε, όταν μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό σύστημα πολιτικών κομμάτων. Δηλαδή θέλουμε να πάμε στην εμβάθυνση της ολοκλήρωσης και να χρησιμοποιήσουμε τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ως δράστες αυτής της ολοκλήρωσης. Ε, είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να εξερευνήσουμε, να συζητήσουμε, γιατί θεωρώ και εντός των τωρινών ευρωπαϊκών πολιτικών κόμματων. Γιατί νομίζω δεν έχει συζητηθεί ακόμα κάτι τέτοια. Δεύτερο, το οποίο αναφέρθηκε νομική βάση. Θεωρώ βασική προϋπόθεση για την πραγματική αναγνώριση και την εντύπωση στη συνείδηση του λαού των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων το να έχουν μια ευρωπαϊκή νομική προσωπικότητα. Δηλαδή θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως υποκείμενα του δικαίου στο, ευρω... στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όχι κάποιος βελγικός μη, κυβερ... μη κερδοσκοπικός σύλλογος, αλλά δομές με νομική υπόσταση. Και αυτό θα έθετε και ένα πλαίσιο να μιλήσουμε για μεταρρύθμιση του εκλογικού δικαίου, του ευρωπαϊκού, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και για ευρωπαϊκά κοινοβούλια στην εθνική σκηνή. Να δούμε βεβαίως και το ζήτημα της επικουρικότητας. Πρέπει να δούμε λοιπόν το συνολικότερο πλαίσιο εδώ πέρα και βεβαίως ανέφερε και ο κ. Σέφνερ ε, ε, τις τρεις φάσεις που υπάρχουν, αδειοδότηση, συμμετοχή σε εκλογές και χρηματοδότηση, είναι πράγματι επίπεδα τα οποία ορίζουν αυτές τις δομές ε, ε, των ευρωπαϊκών κομμάτων ή το πώς θα μπορούσαν να είναι αυτές οι δομές. Τρίτο ζήτημα βεβαίως η συμμετοχή ατόμων. Το πως θα μπορουσαν να ειναι αυτες οι δομες τριτο ζητημα βεβαιω η συμμετοχη ατομων το δικο μας το κόμμα η Ευρωπαϊκή Αριστερά εχθής εξ αρχής έχει μια τέτοια ρήτρα στο καταστατικό Ήδη δηλαδή έχουμε μέλη άτομα, αλλά έχουμε την εμπειρία πως τα κόμματα και, τα ευρωπαϊκά αλλά και τα κόμματα μέλη δυσκολεύονται να ορίσουν τη σχέση ε, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων συλλογικών υποκειμένων ως μελών, δηλαδή των εθνικών κομμάτων και των ατόμων ως μελών. Σε ποιο βαθμό δηλαδή μπορούν να σχηματίσουν την πολιτική, τη θέληση του Ευρωπαϊκού Πολιτικού Κόμματος. Αυτό και στο δικό μας το κόμμα είναι κάτι το ανοιχτό ακόμα που πρέπει να συζητηθεί και θα είναι συναρπαστικό να ακούσουμε εμπειρίες άλλων ευρωπαϊκών ε, κομμάτων, το τι συζητιέται εκεί πέρα, πώς ε, μπορεί να λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Εγώ προσωπικά θεωρώ πως είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση αυτή, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που λένε εγώ θέλω να εμπλακώ στην ευρωπαϊκή πολιτική, όχι στο εθνικό επίπεδο, στο χύψη κόμμα. Είναι κάτι το ε, συναρπαστικό που θα μπορούσε να βοηθήσει στο σχηματισμό των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Τελικό ερώτημα, το οποίο δεν ξέρω, θα πρέπει να παίξει ένα ρόλο στην έκθεση όσον αφορά την δημοσιότητα, το το πώς θα μπορέσουν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να ε, μπορέσουν να δημιουργήσουν θέλετε ένα προφίλ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά και πάλι ξανά στην κάθε χώρα. Πώς δηλαδή η επικοινωνία θα μπορέσει να λάβει χώρα σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις κοινοβουλευτικές ομάδες κτλ. Αυτό είναι αποστολή βεβαίως και των κομμάτων, αλλά νομίζω και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ. Σχεδόν όλοι ξεπέρασαν ε, το χρόνο αγορευσής τους, αλλά παρόλα αυτά δεν ε, ανέπτυξαν το θέμα ιδιαίτερα. Παρά τη Γενική Συμφωνία ότι θα πρέπει τουλάχιστον να εκπροσωπούνται αυτά τα κόμματα από έναν Ευρωβουλευτή. Ο κύριος Νταφ δεν, ήταν, δεν ε, εντάσσεται σε, αυτή, την κατηγορία. Ήταν, όπως πάντα, πολύ ειλικρινής. Είπατε ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα δεν θα πρέπει απλώς να είναι το άθροισμα ή συλλογέ των ε, συνιστοσών τους, των κομμάτων μελών τους. Θα πρέπει να έχουν και μια επιπλέον αξία θέμενη. Ούτε θα πρέπει να περιορίζονται σε, μελέ, ε, σε μέλη ή κόμματα με πανευρωπαϊκή διάσταση. Σε ό,τι αφορά τον κανονισμό του 2004, θα ήθελα να πω ότι το άρθρο 3 με προβληματίζει αφορά τις προϋποθέσεις και το άρθρο 5 τον έλεγχο, την επαλήθευση. Έχω δύο ενστάσεις για την παράγραφο γάμα. μάλλον όχι ως προς τον τύπο, αλλά ως προς την ουσία. Γιατί αν χρησιμοποιηθούν, αν χρησιμοποιηθεί η παράγραφος αυτή ε, που μιλάει για την ε, πολιτική που θα πρέπει να αισθενίζεται τις ευρωπαϊκές αξίες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καταπνίξει ουσιαστικά τους ε, όσους έχουν διαφορετική γνώμη. σε ό,τι αφορά και το θέμα της χρηματοδότησης και αυτά είναι σαν ένα κατάλοιπα του Σοβιετικού Συντάγματος 36. Καλώς, σας ευχαριστώ. Τελευταία παρέμβαση. Ένστεν Στέτερ, εκπρόσωπος της, του Γερμανικού Ιδρύματος για τις Ευρωπαϊκές Μελέτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν εκπροσωπά τα γερμανικά πολιτικά ιδρύματα, αλλά τα, το, το Ευρωπαϊκό Πολιτικό Ίδρυμα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, αλλά εκπροσωπώ και τους συναδέλφους των υπολείπων Ευρωπαϊκών Πολιτικών Ιδρυμάτων. Μετά τον κανονισμό 2002-2003, το 2007 σε ένα παράρτημα ιδρύθηκαν και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα και ο χρόνος έχει δείξει πως η προστιθέμενη αξία θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα μπορούμε να προσφέρουμε αλλά βεβαίως έχουμε και εμείς το ίδιο καθεστώς με τα ευρωπαϊκά κόμματα, γι' αυτό θα ήθελα να πω πως όταν μιλάμε για την αλλαγή, η μεταρρύθμιση του καθεστώτος των ευρωπαϊκών κομμάτων, βεβαίως θα πρέπει να έχουμε και μεταρρύθμιση του καθεστώτος των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων ταυτόχρονα, στο, στο ίδιο πλαίσιο δηλαδή. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου, αυτό θα ήθελα να πω και σε αυτό συμφωνούν μαζί μου και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Ιδρυμάτων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Δεν έχουμε πολύ χρόνο βεβαίως. Λοιπόν, ο πρόεδρος Μάρτιν ζήτησε να μιλήσει. Έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να παρατηρήσω κάποιες αμελιώδεις παρατηρήσεις που έγιναν να απαντήσω σε αυτές. Όσον αφορά τι προτάσει του Γενικού Γραμματέα, συμφωνώ. Και θα ήθελα να τονίσω πώς μιλάμε για μια ουσιαστική βελτίωση αλλά δεν ε, ζητάμε περισσότερα λεφτά. Δεν είναι αυτό το θέμα. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Δεν ζητάν τα κόμματα περισσότερα λεφτά. Απλά υπάρχουν και σημαντικές πρακτικές βελτιώσεις που υπέρχονται. Δεύτερον, η εσωτερική δημοκρατία στο κόμμα μας, εδώ και πολλά χρόνια, λαμβάνουμε αποφάσει κατά πλειοψηφία. Στο συνέδριο και στην πολιτική συνέλευση του κόμματός μας. Οι εκπρόσωποι ορίζονται από τα κόμματα μέλη, τα οποία παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ο καθορισμό του δόγματός μας και του εκλογικού μας προγράμματος. Και όσον αφορά τώρα τα μεμονωμένα μέλη, έχουμε αυτό το οποίο λέμε supporting members, αλλά είμαι διατεθειμένος να δούμε το ζήτημα των μεμονωμένων μελών, τα οποία θα πλαισιώσουν τους εκπροσώπους των ενώσεων μας και των κομμάτων μελών και να έχουν και δικαίωμα ψήφου στο συνέδριο. Αυτό είναι μια σημαντική ανανέωση στην δομή μας που όπως σας είπα λαμβάνει υπόψη κατά πλειοψηφία. Τέλος, για τον πολιτικό ρόλο. Εάν, παραδείγματος χάρη, θέλουμε πανευρωπαϊκή λίστα, στην περίπτωση που θέλουμε να έχουμε πραγματικό ανταγωνισμό στις, Ευρωπα... στις ευρωεκλογές, π.χ. με υποψηφίους ε, στην, για την Προεδρία της Κομισιόν, τότε είναι αναγκαίο τα διάφορα ευρωπαϊκά κόμματα να αποκτήσουν ευρωπαϊκό καθεστώς και νομίζω πως είναι ουσιαστικά αυτά τα οποία διατυπώθηκαν όπως ακούστηκε. Είμαστε αυτή τη στιγμή μη κερδοσκοπικές ενώσεις, διεθνείς ή εθνικές δεν έχουμε ευρωπαϊκό καθεστώς και το χρειαζόμαστε απολύτως όπως λέει και το κείμενο Λάινεν, θα πρέπει να ορίζει δικαιώματα και υποχρεώσεις και να τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα βασισμένη στο ευρωπαϊκό δίκαιο και που θα ισχύει στα κράτη-μέλη. Είναι πάρα πολύ σημαντική μεταρρύθμιση αυτή και χωρίς αυτή τη μεταρρύθμιση τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα δεν θα μπορέσουν να παίξουν τον πολιτικό ρόλο που αναφέρεται στις προτάσεις αυτές, όπως παραδείγματος χάρη την Πανευρωπαϊκή Λίστα, όπως παραδείγματος χάρη την υποβολή υποψηφιωτήτων για τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μόνο με αυτόν τον τρόπο νομίζω μπορούμε να έχουμε περισσότερο αντίκτυπο στη δημόσια στην κοινή γνώμη. Το πρόβλημα και οι δυνατότητες σχετίζονται και με την εμπλοκή βεβαίως των κομμάτων μας. Δεν είναι δυνατόν από ένα κέντρο στις Βρυξέλλες να έχουμε πραγματικό αντίκτυπο στην κοινή γνώμη σε όλες τις χώρες. Πρέπει να ακολουθήσουμε είτε τα μεμονωμένα κόμματα μας, είτε την αυτή δυνατότητα των ατόμων μελών για να έχουμε ένα αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Αυτό μπορεί να γίνει με την ευρωπαϊκή λίστη, με του ανταγωνισμού υποψηφιωτήτων για τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για τις ευρωεκλογές. Με συγχωρείτε, έτσι μίλησα ε, λίγο με πάθο, αλλά αυτά είναι πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στα ευρωπαϊκά κόμματα. Eh, Δεν ζητάω. Αν πάρει κι άλλο το λόγο, παρακαλώ να είστε πάρα πολύ σύντομοι, γιατί μετά θα μείνουμε χωρί διερμηνία. Η κυρία Φρασόνη, πολύ σύντομα πρόεδρε, ευχαριστώ, διότι με το ίδιο πάθο μπορώ να πω ότι συμφωνώ με αυτά που είπε και ο πρόεδρο Μάρτιν μόλι τώρα. Θα ήθελα όμως να πω, απευθυνόμενο προς τον κύριο Τεχρότα, αν κατάλαβα σωστά το όνομα, εάν κάνω λάθος ζητώ συγγνώμη, σχετικά με αυτό που μας είπε όσον αφορά το θέμα του προσωπικού. Είναι απόλυτα θεμελιώδες αυτή τη συζήτηση να κάνουμε μια διάκριση. Το θέμα της αναγνωρίσεως δηλαδή της νομικής του Ευρωπαϊκού Κόμματος από το ζήτημα που καθόρισε την πρώτη μου παρέμβαση σαν γραφειοκρατικό, δηλαδή το καθεστώς του προσωπικού, του staff λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι σε διάφορες περιστάσεις υπήρξαν μάκρος δημιουργικοί για να βρούμε λύσεις επαρκής. Ίσως έχουμε μείνει πίσω. Δεν θεωρώ ότι υπήρξε κάποια τοποθέτηση από πλευρά του Προεδρείου από αυτού, του Κοινοβουλίου. Ε, ο κόσμος το στο Προεδρείο ξέρω ότι έχει θέση υποστήριξη όσον αφορά το θέμα του προσωπικού αλλά απευθύνω μια έκκληση εγώ προς τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών ομάδων να αποφύγουμε να μπούμε σε μια συζήτηση ανταγωνιστική όσον αφορά αυτό το θέμα που θα μας στερούσε για λόγους γραφειοκρατικούς από ένα αμέσο αποφασιστικό για την ταυτότητά μας. Αν και συμφωνώ με αυτό που υπόθηκε από την κυρία Νέιτς, όχι όσον αφορά την νομιμότητα. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα θέμα πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό και κρίσιμο. Όσον αφορά τα ε, mail, τα, τα μεμονωμένα. Και για μας τους είναι περίπλοκο το θέμα, το συζητούμε στο εσωτερικό μας οι κλπ. Για το θέμα συμμετοχής των ατόμων έχουμε ένα δίκτυο υποστηρικτών που ακόμα για να πάρουν την, ε, τα, τα χρήματά σε ποσό τους σχετίζονται με το Εθνικό Κόμμα και αυτό είναι καθοδόν να ξεπεραστεί. Είναι μια διαδικασία που θα γίνει πιο αποτελεσματική όσο πιο χρήσιμο, χρήσιμη μπορούμε να αποδείξουμε ότι είναι δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κόμματο. Κάποιο ομιλητή ρωτήθηκε τι κάνετε στην πραγματικότητα, ποιο είναι ο στόχο. Σίγουρα να κάνουμε χρήσιμα πράγματα, χρήσιμα και ευρωπαϊκά. Συμμετοχή στη συζήτηση, να αλλάξουμε τις απόψεις και να προωθήσουμε θέματα και σε εθνικό και τοπικό επίπεδο που σήμερα δεν έχουν κάποια ε, ευρωπαϊκή χρειά. Για όλα αυτά τα πράγματα χρειαζόμαστε νομικό καθεστώ και επαρκή χρηματοδότηση και να έχουμε υπόψη μα ότι ο στόχος μας δεν είναι να αλλάξουμε σε εθνικό επίπεδο τη συζήτηση, αλλά να ευνοήσουμε την ευρωπαϊκή συζήτηση και μέσω τη συμμετοχή στην εθνική συζήτηση. Ευχαριστώ. Κόρμπε, κύριο Κόρμπε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους ε, βουλευτές που έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Ήταν πολύ χρήσιμο και για μας γιατί ακούσαμε μερικές λαμπρές ιδέες. Θα ήθελα να κάνω μια πρόταση προς την Επιτροπή σας. Δεν θα ήταν σκόπιμο να γίνει μια πιο ευρυθής ανάλυση των εθνικών καταστατικών και καθεστώτων λειτουργίας των κομμάτων. Νομίζω ότι το αναφέρει και η μελέτη του Προεδρίου, Αλλά να δούμε τι είναι αυτό που λειτουργεί καλύτερα. Ποια είναι η βέλτιστη πρακτική σε κάθε κράτο και ως προς τη λειτουργία και ως προς την αναγνώριση του κόμμα, των κομμάτων γιατί ως προς το επίπεδο αναγνώρισης ίσως ε, αντιλήσουμε ενδιαφέροντα στοιχεία από το τι ισχύει στα κράτη. μπορούμε να βρούμε ενδιαφέροντα παραδείγματα και σε εθνικό επίπεδο και για τα θέματα χρηματοδότησης. Γιατί σε πολλές εθνικές νομοθεσίες γίνεται διάκριση μεταξύ της επιστροφής των δαπανών προεκλογικής εκστρατείας και των προϋπολογισμών λειτουργίας. Και εκεί υπάρχει διαφοροποίηση. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιε επιδοτήσει χρησιμοποιούνται για την προεκλογική εκστρατεία, ενώ η αιτήσια χρηματοδότηση σχετίζεται άμεσα με τον αριθμό των ευρωβουλευτών που εξελέγησαν στις τελευταίες ευρωεκλογέ. Και σε ό,τι αφορά τη συγχρηματοδότηση, διαβάσαμε τη μελέτη και βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν ζητούν συγχρηματοδότηση των, των εθνικών πολιτικών κομμάτων. Θα πρέπει λοιπόν να το εξετάσουμε για να εξασφαλίσουμε ισότητα όλων των κομμάτων απέναντι στη χρηματοδότηση. Και νομίζω ότι η αρχική πρόταση του Γενικού Γραμματέως για την ε, κατάργηση των τοπικών ε, χρηματοδοτήσεων είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές είχαν ε, πολύ μακροσκελή συζήτηση για τα άμεσα μέλη όχι και για να αποφύγουμε αντιπαράθεση μεταξύ των εθνικών και των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, κρίναμε σκόπιμο όλα τα, ότι όλα τα μέλη των εθνικών κομμάτων θεωρούνταν ω μέλη του Ευρωπαϊκού Πολιτικού Κόμματος. Μόνο όμω όσοι το επιθυμούν μπορούν να γίνουν ε, ενεργά μέλη, στρατευμένα μέλη κατά κάποιο τρόπο του Ευρωπαϊκού ε, Σοσιαλιστικού Κόμματο, που είναι πιο δραστήρια, έχουν πιο ακτιβιστικό ρόλο. Δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο και για το ΕΛ και για τα άλλα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Νομίζω ότι περισσότερα ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο. Για να αποφύγουμε ανταγωνισμό μεταξύ των εθνικών και των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα επιπλέον επίπεδο δραστηριοτήτων για τα μέλη μας. Και φυσικά έχουμε και ένα τμήμα τοπική συμμετοχή, όπω συμβαίνει και για του αρχηγού των εθνικών κομμάτων. Στείλαμε και γραπτό στι απαντήσει μα στο ερωτηματολόγιο τη συζήτηρια για να εμπλουτίσουμε και εμεί με τη συμβολή μα στη συζήτηση. Κυρία Νέιτ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ συνάδελφε, σα εκπλήσει το ότι επειδή είμαι φιλελεύθερη, ε, φρύτη ακούγοντας κάποια από τα πράγματα που υπόθηκαν που θέλουν να διοργανώσουν κάθε μικρή λεπτομέρεια της δημιουργίας, της λειτουργίας και της εσωτερικής διοργανώσεως όχι μόνο των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, αλλά και ενδεχομένω και των εθνικών πολιτικών κομμάτων. Εκεί νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ μακριά. Πραγματικά πιστεύω ότι πάμε πολύ μακριά. Θα πρέπει να αφήσουμε περιθώριο και χώρο σε ατομικέ πρωτοβουλίες, σε πρωτοβουλίες μικρών ομάδων που θέλουν να μπουν στην πολιτική περιπέτεια, χωρί ε, από την αρχή να πρέπει να φροντίσουν για να γίνουν αποδεκτοί για να συμμετάσχουν στην πολιτική ζωή της χώρας τους. Εκεί νομίζω ότι ξεπερνάμε κάποια όρια και πηγαίνουμε πολύ μακριά και θα μπορούσαμε να παρασυρθούμε ίσως, να προσπαθήσουμε να στριμώξουμε τη δημοκρατία για το καλό της βέβαια και να μετακινηθεί πολιτικός αυθορμητισμός σε άλλες σφαίρες, σε άλλους τόπους ε, και νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να αποφύγουμε. Τούτων λεχθέντων θα ήθελα να κάνω άλλο ένα σχόλιο που δίνει μια συνέχεια σε αυτά που είπε ο Wilfried Martens. Δηλαδή αδιαμφισβήτητα εντός των ευρωπαϊκών πολιτικών μας κομμάτων υπάρχει μια τάση αδιαμφισβήτητη, μια ένταση μάλλον μεταξύ των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των δομών τους και των εθνικών κομμάτων. Υπάρχει μια ένταση δεν υπάρχει ε, ταυτότητα απόψεων πάντα, ούτε υπάρχουν κοινά συμφέροντα. Και για να φροντίσουμε ούτω ώστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μπορούμε να συνεχίσουμε να θα από αυτά που ζουν τα κόμματα μέλη μας, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις ευαισθησίες τους, αυτά που σκέφτονται, να προσπαθούμε να τα προσελκύσουμε και να προσχωρήσουν. τα πολιτικά προγράμματα τα περιορισμένα που ετοιμάσαμε κατά τη διάρκεια δύο ετών εν ώψη των ευρωπαϊκών εκλογών που προηγήθησαν και το πρώτο από ήμασταν, ήταν το πρώτο που ομόφωνα ειδητήθηκε από το 1976 από το συνέδριό μας. Όλα τα προηγούμενα προγράμματα ε, απερίφθησαν ε, από ένα ή περισσότερα από τα κόμματα μας και χρειάστηκε να γίνει προσπάθεια ε, να τα πείσουμε. Και απευθύνω μια έκκληση προς τους συναδέλφους της ε, Συνταγματικής Επιτροπής. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το ότι τα εθνικά κόμματα δεν είναι ακόμα όλα πεπισμένα για τη χρησιμότητα ή το εφικτόν ή τον πρακτικό χαρακτήρα ε, των εθνικών φορέων. Χρειάζεται ενημέρωση, χρειάζεται πειθό αν δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε άρνηση όσον αφορά αυτή την περιπέτεια στην οποία θέλουμε να προχωρήσουμε, που θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά που θα πρέπει να τύχει τη υποστήριξης και της προσχωρήσεως των εθνικών μας κομμάτων. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο κύριος Λοράνκη, παρακαλώ να είναι σύντομο. Ένα σχόλιο συμπληρωματικό όσον αφορά τις ατομικέ, ε, τι ε, ατομικές, τις άμεσες Είναι ένα σύστημα που εξετάσαμε, αλλά που δημιουργεί προβλήματα που αναφέρθηκαν ποικιλοτρόπως. Δηλαδή, σχέσεις μεταξύ των αμέσων μελών και των κομμάτων μελών, αλλά θα ήθελα να κάνω ένα πολιτικό σχόλιο σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Νταφ, που συνέδε αυτό το θέμα με τη δυνατότητα της, ε, της υπερεθνικής λίστας. Αν θα μπορεί να γίνει μετά εθνική δημοκρατία να υπάρξει κανένα σύστημα, κατά την άποψή μου, δεν θα εξαλείψει το πρόβλημα της δημοκρατικής οικοδόμησης των στόχων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δεν αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα ε, επικοινωνίας και ας υπάρχει. Και η συζήτηση που γίνεται στην Ευρώπη με τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά πολύ πιο σοβαρά πράγματα. Νομίζω λοιπόν ότι οι προσπάθειες που πρέπει να καταβάλουμε θα πρέπει να έχουν σαν στόχο την ποιότητα της δημοκρατικής συζήτησης, στη συνέπειες πολιτικής συζήτησης όσον αφορά τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Δεν θέλουμε να το ξεπεράσουμε αυτό. Δεν θέλουμε να υπερκεράσουμε τις αντιφάσεις που βλέπουμε σήμερα χωρίς να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή πολιτική ε, γνώμη όσον αφορά τους στόχους του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Είναι θεμελιώδες θέμα αυτό, το περιεχόμενο δηλαδή του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ο τελευταίος που ζήτησε το λόγο είναι ο συνάδελφος Νταφ. Παρακαλώ, είστε σύντομος. Η συγγήτρια μπορεί ίσως να δώσει κάποιες απαντήσεις το απόγευμα να απαντήσει. Όχι τώρα, το βράδυ, έτσι. Το απόγευμα. Ο κύριος Νταφ. Υπάρχουν εντάσεις και τάσεις μεταξύ των εθνικών πολιτικών δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των ε, ομοσπονδιακών συστημάτων. Αυτό είναι φυσικό ε, το ευρωπαϊκό σύστημα. Δεν πρέπει να σε εκπλήσει αυτό. Σίγουρα δεν νομίζω ότι θα πρέπει να τρομάζουμε ε, όσον αφορά το ότι υπάρχει ένα στοιχείο ανταγωνισμού μεταξύ των υπερεθνικών ή των μεταεθνικών πολιτικών δυνάμεων ε, που διαμορφώνονται και των παλιών εθνικών πολιτικών δυνάμεων. Είναι καλό για την πολιτική να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ διαφόρων επιπέδων διακυβερνήσεως, όπως συμβαίνει και στην οικονομική σφαίρα, και έχουμε μεγάλη εμπειρία οικονομικής ολοκληρώσεως. Δεν είχαμε επαρκή εμπειρία όσον αφορά τη δημοκρατική ολοκλήρωση μέχρι τώρα. Για να το ξεκαθαρίσω, προτείνω ότι θα έπρεπε να αποτελέσει κριτήριο για την διαμόρφωση ενός Ευρωπαϊκού Πολιτικού Κόμματος με συγκεκριμένο καθεστώς ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα τμήμα ξεχωριστό πολιτών. Δεν θέλουμε να εξαιρέσουμε ε, τις εθνικές συνιστώσεις που βεβαίως θα εξακολουθούν να αποτελούν τον πυρήνα, την καρδιά, το βασικό σώμα των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, αλλά θα πρέπει να συμπληρώνονται από την διαμόρφωση ενός τμήματος πολιτών, το οποίο τμήμα θα έχει συγκεκριμένα θεσπισμένα δικαιώματα όσον αφορά το δημοκρατικό διακομματικό σύστημα των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Και επίσης θα ήθελα να προσθεθεί και το εξής. Ότι στα τμήμα των προτάσεων για ένα υπερεθνικό εκλογικό σύστημα να δημιουργηθεί μια εκλογική αρχή ευρωπαϊκή που θα πρέπει να ρυθμίζει τη διεξαγωγή αυτού του τμήματος των εκλογών. Σα ευχαριστώ. Θεωρώ ότι η πρωινή συνεδρίαση υπήρξε πάρα πολύ πλούσια και τα σημεία θα, που αναφέρθηκαν θα πρέπει ε, να ίσως συμπεριληφθούν μέσω γραπτών συνεισφορών που αποσταλούν ε, και αναγκαίες από κάποιους από εσά. Θα επαναλάβουμε τις εργασίες μας το απόγευμα. Θα δώσουν περισσότερο περιθώριο από αυτό που προβλεπόταν. Στις 3 και 4 Παρακαλώ όμω να είσαστε ακριβεί, να είσαστε εδώ. 3 και τέταρτο. Θα μπορούσα να πω να ξεκινήσουμε στι 3, να ξεκινήσουμε πραγματικά στι 3 και τέταρτο, αλλά παρακαλώ λέμε 3 και 4, είστε εδώ 3 και 4, διότι έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλου του εκπροσώπου των Ευρωπαϊκών Κομμάτων. Διακόπη τη συνεδρία σα. Καλή σα όρεξη.